Συνεχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Θα σας καλωσορίζω στην απογευματινή συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Θα συζητήσουμε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus. Και θα δώσω μέσω στο λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Λόπε Φοντανιέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους και εσάς μετά τις διακοπές που ελπίζω να ξεκουραστήκατε, να τις χαρήκατε και να μπορέσουμε ξανά να στρωθούμε στη δουλειά με κουράγιο και δύναμη για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή πριν το τέλος της θητείας, ελπίζω. Ας το προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Πριν ε, αρχίσω να σας μιλώ για το σχέδιο και τις τροπολογίες στη συζήτηση, θέλω να σας πω ότι γενικά συμφωνώ με τα όσα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το είπα και την περασμένη φορά πριν τις στενές διακοπές και ιδιαίτερα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, συγχωνευτούν διάφορα ταμεία για να έχουμε και συνέργειες αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία. Όπως προτείνεται να συνδέονται περισσότερο με τις ειδικέ συστάσεις αναχώρα τα ταμεία αυτά και με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Αυτά τα δύο αρχικά ε, είναι πολύ σημαντικά. Όπως είπα πριν το θέρος, η έκθεση μου καλύπτει τα σημαντικότερα σημεία όπως και οι τροπολογίες ε, στο ίδιο κλίμα και στο ίδιο πνεύμα του κειμένου. Χρόνο δεν έχουμε, είναι πολύ περιορισμένος και αν θέλουμε να βγάλουμε καλή έκθεση που θα συνεισφέρει στη βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής κατάστασης αλλά και με μεγαλύτερη ε, υποστήριξη και πλειοψηφία πρέπει να εργαστούμε από κοινού. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό ε, σήμερα να ακούσω εσάς όλες τις γνώμες, τις παρατηρήσεις και τις ανησυχίες και τις αντιρρήσεις όλων των συναδέλφων. Ακόμα είναι πολλές οι προκλήσεις, οι κοινωνικές και οι εργασιακές, στις οποίες οφείλει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η ενεργεία των νέων, η μεγάλη ε, επισφάλεια ε, ε, οι μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες ε, ευρωπαϊκές περιφέρειες καθώς και ο μεγάλος αριθμός νέων που είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και άσκησης. Στο μελλοντικό λοιπόν Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus ενισχύεται η κοινωνική διάσταση και οι στόχοι της. Είναι αυτό καλή είδηση για όλους αν καταφέρουμε να φέρουμε σε αίσιο πέρας αυτή την προσπάθεια. Όπως σας είπα και προηγουμένως για όλα αυτά θεωρώ πολύ σημαντικό να συγχωνευθούν τα διάφορα ταμεία στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus γιατί αυτό ε, θα βελτιώσει τη λειτουργία του, την πρόσβαση για τους δικαιούχους και θα έχουμε και συνέργειες ακριβώς επειδή θα είναι πιο εστιασμένη όλη αυτή η προσπάθεια. Για τους νέους ιδιαίτερα. Θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ ψηλή νεανική ανεργία και εμείς το γνωρίζουμε εδώ, είναι διπλάσια από το συνολικό ποσοστό ανεργίας. Ε, η μη συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας δεν είναι μόνο εις βάρος της κοινωνικής συνοχής στην Ένωση αλλά είναι και μια απειλή για την ίδια την βιωσιμότητα του κράτους ε, ε, πρόνοιας η πρωτοβουλία για την ε, απασχόληση των νέων ήταν πολύ σημαντική για την προώθηση των νέων στην αγορά εργασίας. Οι χώρες που έχουν την περισσότερη νεανική ανεργία γενικά είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν και περισσότερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Και γι' αυτό το λόγο θα προτείνω 10 με 15% αύξηση των πόρων ε, για την απασχόληση των νέων, 15 με 19 ε, τον των νέων που δεν είναι σε κατάρτιση, εκπαίδευση, ε, μαθητεία ή ε, απασχόληση. Επίσης, η φτώχεια συνδέεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό και θέλω να επιμείνω σε αυτό. Θεωρώ θετικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να δώσει το 25% των πόρων στο στόχο αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι αρκεί αυτό το ποσοστό. Ξέρω ότι είναι περιορισμένοι οι πόροι και τα χρήματα, αλλά με ένα 25% νομίζω δεν καλύπτεται. Θα πρέπει να έχουμε ένα 2% επιπλέον για να καλύπτουμε τις βασικές ε, διατροφικές ανάγκες και τις πρώτες ανάγκες ε, των πιο απόρων. Η επιστημιστική βοήθεια προς τους απόρους είναι πολύ σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταπολεμάει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ξέρω ότι μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα η πολιτική των κρατών, ε, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό επίσης σημαντικό να προωθήσουμε την ενεργό συμμετοχή των ε, ΜΚΟ, ε, ιδίως εκείνων που συνεργάζονται με την κοινότητα των Ρωμά, αλλά και με ανθρώπους που ε, ζουν στη φτώχεια γιατί χρειάζονται ειδικά προγράμματα. Και πάντα να είναι τα προγράμματα σχεδιασμένα με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το Ταμείο θα πρέπει να προωθεί την ισότητα των ευκαιριών και τη μη διάκριση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση και τη διατήρηση και την προώθηση της αγοράς εργασίας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χάσματα ακόμα και διαφορές ε, μεταξύ των περιφερειών αλλά και στο εσωτερικό των περιφερειών. Για να έχουμε ενιαία ανάπτυξη λοιπόν χρειάζεται τριπλή προσέγγιση, οικονομική, κοινωνική αλλά και εδαφική. Η Ήπεθρος και οι περιοχές αυτές που έχουν ε, προβλήματα σοβαρά δημογραφικά αλλά και γεωγραφικά και μετρολογικά έχουν και τις λιγότερες ευκαιρίες και τις λιγότερες υποδομές. Δεν φτάνει που έχουν μεγάλα προβλήματα και γύρανση στο πληθυσμό. Αν ξεχάσουμε λοιπόν αυτές τις ιδιαιτερότητες της υπαίθρου και της περιφέρειας, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε στους στόχους που προτείνονται. Αυτά κυρία Πρόεδρε είναι τα βασικά των προτάσεών μου που έχω βάλει στο πρώτο προσχέδιο έκθεσης που όπως σας είπα και πριν το καλοκαίρι θα το εμπλουτίσω με τροπολογίες που θα πηγαίνουν στη διακατεύθυνση φυσικά με την έκθεσή μου. Αυτά. Σταματώ εδώ την ανάγνωση. Είμαι στη διάθεσή σα και ελπίζω να μπορέσουμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε το σύντομότερο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much for that. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγική σας αυτή παρέμβαση. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τους κοιόδης συγητές. Ο κύριος ε, Μπράντο Μπενιφέ έχει πρώτος το λόγο από την Ιταλία, από την ομάδα των Σελιστών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη συνάδελφο Βερόνικα Λόπε Φοντανιέ για την παρουσίαση αυτή του σχεδίου έκθεσης. Εξ αρχής θα πρέπει να πω ότι πολλά από τα σημεία τα οποία έθιξε η συγγήτρια με βρίσκουν σύμφωνο. Είμαι και εγώ πεπισμένος ότι θα καταφέρουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια κοινή και γρήγορη εργασία για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μας περιορίζει πολύ όμως ο χρόνος. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση που έχει να κάνει με τις επερχόμενες ευρωεκλογές. Επομένως θα πρέπει και για την πρόταση αυτή αλλά και για πολλές άλλες προτάσεις να εργαστούμε πολύ σκληρά και πολύ γρήγορα και από τεχνική, αλλά και πολιτική πλευρά, καθώ το ζήτημα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτική πλευρά. Εμεί, ω σοσιαλιστέ, είμαστε πεπισμένοι θα καταφέρουμε συνεργαζόμενοι με την κυρία Λόπε Φοντανιέ να καταλήξουμε σε μια φιλόδοξη κοινή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να καταλήξουμε και σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο. Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω κάποια σημεία τα οποία θεωρώ ότι είναι κέρια σημασία και τα οποία ουσιαστικά θα αποτελέσουν και το αντικείμενο των τροπολογιών που θα καταθέσω. Θεωρώ ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και θα πρέπει να φτάσει πραγματικά σε αυτού που το έχουν περισσότερο ανάγκη, στι πιο μειονεκτούσε δηλαδή ομάδε. Θα πρέπει να λύσουμε λοιπόν διδάγματα από την εφαρμογή του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να καταφέρουμε να επιφέρουμε τι απαραίτητε βελτιώσει και διορθώσει. Πρώτα απ' όλα να καταφέρουμε να απλουστεύσουμε τη διαχείριση του προγράμματο. Θα πρέπει αυτό να αποτελεί κοινό μα στόχο, να καταφέρουμε δηλαδή να απορροφήσουμε περισσότερου πόρου και να καταστήσουμε τα προγράμματα πιο αποτελεσματικά. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus θα πρέπει να προσαρμόζεται στι τοπικέ ιδιαιτερότητε, θα πρέπει να συνάδει με τα υπόλοιπα προγράμματα και ταμεία, θα πρέπει να γίνεται πιο αποτελεσματικό, αλλά και λιγότερο γραφειοκρατικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απλοποιηθούν οι κανόνες για όλους του εμπλεκόμενου φορεί. Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν περισσότερο την έννοια τη εταιρική σχέση και να κινηθούμε εδώ πέρα στο δρόμο που έχει δείξει στην έκθεση αυτή η συγγήτρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να καταφέρουμε να τονίσουμε περισσότερο την εδαφική διάσταση του Ταμείου αυτού, να καταφέρουμε να εμπλέξουμε περισσότερο τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ, του κοινωνικού εταίρου, καθώ επίση και την κοινωνία των πολιτών, στην όλη αρχιτεκτονική των προγραμμάτων, αλλά επίση και στην εφαρμογή του, την επιθεώρηση και τον έλεγχό του. Προτείνεται επίση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus να συντονιστεί περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ιδίω με τι ειδικέ αναχώρα συστάσει και με τι βασικέ αρχέ του κοινωνικού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Θεωρώ ότι η προσέγγιση αυτή είναι απόλυτα λογική. Πιστεύω ότι όντως θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε μία προσέγγιση η οποία θα οδηγήσει σε περισσότερες οικονομίες αλλά και σε καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τις κοινωνικές πολιτικές και την πολιτική συνοχής. Ας καταφέρουμε όμως να προσπίσουμε στο κείμενο αυτό τη βασική αρχή που το διέπει, δηλαδή ότι θα πρέπει πραγματικά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δικαιούχων και να είναι ευπροσάρμοστο στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες και να μην γίνει ακόμα ένα άκαμπτο νέο μέσο, νέο εργαλείο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αντίθετα, νομίζω ότι θα πρέπει να προωθεί περισσότερο τις κοινωνικές ανάγκες και να προσαρμόζεται πραγματικά σε αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus θα πρέπει επίσης να συνάδει περισσότερο με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα και θα πρέπει επίσης να μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τελικά ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο πιο κοινωνικό αν θέλετε. Προκειμένου προκειμένου το πετύχουμε αυτό, πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένους δείκτες, καθώς επίσης και το κοινωνικό scoreboard, το κοινωνικό πίνακα αποτελεσμάτων. Θα μπορούσα να παραθέσω πολλά περισσότερα επιχειρήματα, αλλά προτιμώ να ολοκληρώσω στο σημείο αυτό, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιαστούμε και στο εξή σημείο, στην εγγύηση για τους νέους. Ξέρετε ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ουσιαστικά ενσωματώνεται και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε μέσω του νέου κοινωνικού αυτού ταμείου να προωθήσουμε τι πρωτοβουλίε αυτέ για την απασχόληση των νέων σε τοπικό επίπεδο, να καταπολεμήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την ανεργία των νέων και να καταφέρουμε να έχουμε και ένα καλύτερο συντονισμό διοικητικό και διαχειριστικό. Μα δίνεται επίση μέσω του νέου αυτού ταμείου δυνατότητα να ενισχύσουμε την εγγύηση για του νέου, να καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε την όλη εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει τελευταία χρόνια. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε πραγματικά να θέσουμε ω προτεραιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση την καταπολέμηση τη ανεργία των νέων, έχοντα απαραίτητου πόρου και τα απαραίτητα μέτρα τα οποία θα δημιουργήσουν νέε θέσει απασχόληση. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να συγκεράσουμε την απασχόληση με τι υγειονομικέ υπηρεσίε, τι υπηρεσίε για την κοινωνική στέγαση και τι υπόλοιπε κοινωνικές υπηρεσίες. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και βλέπω σε μια θετική συνεργασία με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπου συναδέλφου. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you. Then I'll give the floor to ε, Και εμεί σα ευχαριστούμε. Η κυρία Ολυρίκη Τρεμπέσιου τώρα έχει το λόγο εξ ονόματο του ECR. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία εισηγήτρια, κυρία Λόπε Φοντανιέ η πρότασή σας, όπως είπατε και εσείς η ίδια, προσανατολίζεται σε γενικές γραμμές ε, στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μια έκθεση που αφορά κυρίως την αναδιάρθρωση των οργανισμών ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλό είναι αυτό και το θεωρώ και εγώ και ομάδα μου λογικό. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει την ελευθερία στο μέλλον να οργανώνεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα ελπίζουμε και με πιο διαφανείς διαδικασίες για τους πολίτες και για την οικονομία. Δυσκολεύουν τα πράγματα εκεί όπου τα οικονομικά μέσα θα πρέπει να αλλάξουν προορισμό ή που ε, το πεδίο ε, χειρισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διευρύνεται για να κατανέμει τα κονδύλια με τρόπο λέει πιο ευέλικτο ε, και ε, σε προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ήδη έχει απειλήσει ο πρόεδρος Γιούγκερ ότι ε, θα δοθούν λιγότερα χρήματα στο μέλλον σε ισχυρά κράτη όπως είναι η Γερμανία και μένα έχουν ανάψει τα λαμπάκια και χτυπάνε τα καμπανάκια γιατί προβλήματα έχουν και τα πιο πλούσια κράτη στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να δεχτούμε μείωση των επενδύσεων γιατί λέει για να διατηρηθεί το ευρώ πρέπει να στείλουμε περισσότερα λεφτά στην Νότια Ευρώπη. Υπάρχουν σε πολλές χώρες προβλήματα που δεν υπάρχουν κρατικές δομές ή δεν λειτουργούν σωστά και τα χρήματα δεν πιάνουν τόπο και δαπανώνται ε, απλώς και μόνο επειδή είναι ευρωπαϊκά κράτη αυτά τα κράτη. Ενώ στη Γερμανία και στην Αυστρία έχουμε προγράμματα που τρέχουν και λειτουργούν καλά και δεν βλέπω το λόγο να τα περικόπτουμε. Χαίρομαι για την τροπολογία 3 της εισηγήτριας που τονίζει τα ειδικά μελήματα ε, και τα θέματα των ταμείων ε, δεν θα πρέπει να αλλάξουν, λέτε, ε, και θέλουμε να την συμπληρώσουμε αυτή την τροπολογία, να συνεχίσουν να δαπανώνται τα κονδύλια εκεί που πιάνουν τόπο και όλες οι περιφέρειες καταρχήν να παραμένουν επιλέξιμες. Γι' αυτό θεωρώ όλο και πιο προβληματικό ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιούνται λέει, στο μέλλον για να εντάσσονται ε, στην κοινωνία μας περισσότερο πολίτες τρίτων κρατών, όπως λέει η τροπολογία 1. Διαφωνώ για τη μετανάστευση. Υπάρχουν άλλα ταμεία για το άσυλο και τη μετανάστευση. Υπάρχει ειδικό εργαλείο εκεί. Εάν το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη θέλουν περισσότερα χρήματα προς τα εκεί, να πάνε να τα ζητήσουν από το συγκεκριμένο ταμείο με ε, ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Κατά τα άλλα θα πρέπει να αφήνουμε στα χέρια των κρατών μελών πόσους μετανάστες μπορούν να υποδεχτούν και πόσα χρήματα θα διαθέσουν για την ένταξή τους. Και η προθυμία των κρατών ε, είναι περιορισμένη, αλλά περιορισμένα είναι και τα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα πρέπει να παραφορτώνουμε τώρα εδώ ε, τα ταμεία και να αναμειγνύουμε με ε, άλλα ταμεία και με άλλες ανάγκες και απαιτήσει. Θα κάνουμε σχετικά τροπολογίες και χαίρομαι για τη γόνιμη συνεργασία που σίγουρα θα έχουμε με την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ε, now... Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Σελίμοβιτς, εκ μέρους της ομάδας Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να πω ότι στηρίζουμε πολύ θερμά ε, το θέμα ότι ε, έχουν συγχωνευτεί όλα τα διάφορα ταμεία. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο και να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων που παραμένει σε απαράδεκτα ψηλά επίπεδα σε κάποια κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να αναφερθούμε και στις δημογραφικές αλλαγές και ιδιαίτερα μου αρέσει η αναφορά στην ανάγκη ε, συμπερίληψης ε, των μεταναστών, γιατί ξέρουμε ότι κάποιες χώρες έχουν ε, καταβάλει περισσότερες προσπάθειες από άλλες στην πρόσφατη μεταναστευτική κρίση. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι θα πρέπει να υποδείξω ορισμένα σημεία. Η Οι από κέντρες περιοχές ε, είναι, χρειάζονται κυρίως τις υποδομές. Δεν αναμένω από το ESF συν να αντικαταστήσει αυτή την κατάσταση. Δεύτερον, συρίζω αυτό που έχει γραφτεί στην έκθεση και εδώ σχετικά με την ανάγκη ε, να προσαρμόσουμε αυτό το μείωση στη νέα ε, κατάσταση μετά το Brexit. Η συμπερίληψη των ΜΚΟ χρειάζεται, θα πρέπει να διαβελευτούμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, διότι αυτές θα επηρεαστούν και θα είναι οι δικαιούχοι αυτών των ταμείων. Επίση, χώρες με ψηλές ομάδες needs ε, θα πρέπει να υποστηριχθούν, ε, θα πρέπει να ε, καταβληθούν περισσότεροι πόροι για να στοχεύσουμε δράσεις ιδιαίτερα για αυτές τις ομάδες νέων. Η συγκέντρια αναφέρθηκε στο 15%, θα πρέπει να το αυξήσουμε ίσως και περισσότερο. Επίσης, ηλική στήριξη. Θα πρέπει να έχουμε ε, υποστηρικτικά μέτρα χωρίς αποκλεισμούς, διότι ένα ε, δάνειο δεν λύνει τα προβλήματα μακροπρόθεσμα. Ε, αν δεν συμπληρώνεται με άλλα μέτρα, θα είναι μόνο μια βραχυπρόθεσμη λύση η παροχή επιστηστικής βοήθειας και μόνο. Θα πρέπει να δούμε πώς αλλάζουν οι προτεραιότητές μας και πώς ε, μπορούμε να ε, καταπολεμήσουμε τα προβλήματα. Ο διοικητικό φόρτος θα πρέπει να είναι στο ελάχιστο, θα ε, πρέπει να μην προσεθούν επιπρόσθετα προβλήματα διοικητικά σε, ορισμένε περιπτώσει υπάρχει τόσο μεγάλο φόρτο που τελικά ε, καταβάλλονται προσπάθειε περισσότερο ε, για, και τα χρήματα καταβάλλονται περισσότερο για αυτό. Θα, ε, οι ανάγκε κατά χώρα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα και του στόχου που έχουν επιτευχθεί. Αυτέ θα είναι οι προτεραιότητε στην δυνατότητα απορρόφηση των πόρων τέλος. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων είναι θέμα ανησυχία, διότι ε, σε μερικές περιπτώσεις δεν έχουμε τα αποτελέσματα που ελπίζαμε. Σε άλλες περιπτώσεις είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα πρέπει να συγχωνευτεί μέσα στο ESFC, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα την αξιολόγηση του γιατί ε, σε κάποιες χώρες υπήρχε επιτυχία και σε άλλες όχι για να δούμε πώς να γίνει η συγχώνευση και να ε, καταβληθούν αυτά τα ποσά ε, καταλήλως. Θα υποβάλουμε τροπολογίες σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για την παράταση της προθεσμίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Τσίμερ ε, που εκπροσωπεί την ομάδα Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της και τις ε, τροπολογίες. Ε, θεωρώ καλό ε, αυτό που είπε για τη βασική κατεύθυνση της έκθεσης μπορούμε και εμείς να την υποστηρίξουμε και τονίζω ότι η καταπολέμηση της ένδυας και της φτώχειας είναι εξαιρετικό. Επίσης υποστηρίζω και το στόχο ε, να συμπληρωθεί το 25% για ε, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τα χρήματα που πηγαίνουν στην καταπολέμηση της ακραίας στόχιας και την ενίσχυση της αρχής της εταιρικής σχέσης και με την ε, αντίστοιχη ρύθμιση του κώδικα δεοντολογίας. Λοιπόν, προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε και θα συνεργαστούμε μαζί σας με μεγάλη χαρά και με τους υπόλοιπους και ηγητές. Θα ήθελα όμως να προσθέσω και κάποιες επιπλέον θέσεις μας για να σας δείξω και προς τα που θα κινηθούν οι δικές μας τροπολογίες. Πρώτον, στους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο άρθρο 4 θέλουμε να τονιστεί ότι εδώ πρόκειται για πρόσβαση σε απασχόληση υψηλής ποιότητας. Όχι μια απασχόληση και ότι να είναι και επισφαλής και δεν πειράζει. Όχι, αυτά θέλουμε να τα αποφύγουμε. Ε, όχι μόνο με τα διορθωτικά ταμεία να τα στηρίξουμε, αλλά γενικότερα. Ε, επίσης μας ενδιαφέρει και θεωρούμε σημαντικό να υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να ε, έχουν ένα προεπολογισμό που να λαμβάνει υπόψη του το φύλλο με ειδικούς στόχους και επίσης σε σχέση με αυτό που είπατε εσείς για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού είπατε τουλάχιστον 30% το τουλάχιστον με βρίσκει σύμφωνη. Μήπως να πούμε και περισσότερο. Για την κοινωνική ένταξη. Και σε ό,τι αφορά από εκεί και πέρα ε, τους απόρους και την ηλική του στήριξη Βεβαίω και αυτό θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον 4% για να, να φτάνει στο 4% για να μην πω στο 5% του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού ε, Κοινωνικού Ταμείου. Και μάλιστα θέλουμε επιπλέον χρηματοδότηση. Και η συγχρηματοδότηση είναι 85% ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε αυτά τα θέματα της ακραίας φτώχειας και των απόρων. Να μην μειωθεί γιατί είναι τα μοναδικά προγράμματα που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη, ενώ οι ανάγκε είναι τεράστιες και θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι για εκείνους που έχουν πρόβλημα. Συμφωνώ πολύ με τον αδερφό από τους φιλελευθέρους να έχει συνεχιστεί η βοήθεια προς τους απόρους και η ηλική και η επιστηστική. Και όταν δίνονται αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να είναι εγγυημένη και η συνέχιση της βοήθειας γιατί στα τρόφιμα αυτή είναι συνήθως έκτακτη επίγουσα επισητιστική βοήθεια, ενώ αυτό που χρειάζεται είναι στρατηγική υποστήριξη και ε, ένταξη των ανθρώπων αυτών. Για την Επιτροπή ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ, είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, που υπάρχουν και πολλές και ποικίλε εξακολουθούμε να το υποστηρίζουμε και καλό θα ήταν να το κάνουμε και στο μέλλον. Και για τους δείκτες να πω δύο λόγια, ιδιαίτερα τους δείκτες του output θα πρέπει από την αρχή να ε, απλουστευθούν. Και η συλλογή στοιχείων για το τελικό δικαιούχο θα πρέπει να είναι προαιρετική. Δηλαδή, να μην εξαρτήσουμε τίποτα από την προθυμία κάποιου να δίνει πληροφορίε και δεδομένα ε, και να μην του περικόψουμε προφανώς τη βοήθεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοτομείο ΣΥΝ θα πρέπει να μπει και στη συζήτηση που κάνουμε ταυτόχρονα για ε, το γενικότερο κανονισμό για τα διαρθωτικά ταμεία. Για μένα είναι προβληματικό το άρθρο 10 η μεταφορά πόρων από το ε, ESF Plus στο Invest EU. Ξέρουμε ότι το επενδύστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, InvestEU, είναι ένα εργαλείο για την αγορά ε, και πρόκειται κυρίως για κέρδη από την αγορά και όχι για κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θέλουμε να πάρουν λεφτά από το κοινωνικό ταμείο για να το πάνε στις επενδύσεις. Αυτό θα ήταν ε, κατά των προθέσεων και των σκοπών ε, αυτών των πόρων. Επανειλημμένα έχουμε πει εμείς ότι είμαστε κατά της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω. ότι η σύνδεση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΣΥΝ με το κοινωνικό εξάμενο ε, σημαίνει συγκέντρωση ε, σε εθνικό επίπεδο και πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε και πώς θα μπορέσουμε να προβλέψουμε την καταπολέμηση περιφερειακών διαφορών στα κράτη-μέλη, δηλαδή μεταξύ των περιφερειών και να λαμβάνονται υπόψη ε, οι τοπικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ε, οι διάφορες ανάγκες που έχουν και ε, απαιτήσει. Να μην είναι όλα αυτά κεντρικά από την κεντρική κυβέρνηση και μετά να μοιράζονται κατά μέσο όρο ερήμην των ενδιαφερομένων. Προσφέρουμε λοιπόν την υποστήριξή μας, θα κάνουμε τροπολογίες και ε, προσβλέπω σε μια αγαστή όσο και ταχεία συνεργασία. Ευχαριστώ. Thank you. Then I'll give the floor to ε, Madam Reinke, representing the Greens. The floor is yours. Κυρία Ράινκε, έχει το λόγο. Συνόματος των Πρασίνων, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Το είπε και η εισηγήτρια και πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε πολλά σημαντικά ζητήματα θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, δεν θα μακρηγορήσω, πάντως οι προσδοκίες μας είναι ιδιαίτερα υψηλές, γιατί η ανάλυση καταδεικνύει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σαφώς, σαφές πρόβλημα με τις όλο και αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες, ιδιαίτερα εκτεταμένες και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ας μην το ξεχνάμε, είναι από τα βασικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε, να περιορίσουμε αυτές τις ανισότητε Άρα ασκείται σε εμά πίεση για να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Θα ξεκινήσω με κάτι που ήδη υπόθηκε, το πώς μπορούμε να συνδέσουμε, το Μπράντο Μπενιφέ αυτό, να συνδέσουμε το ταμείο αυτό με τον κοινωνικό πυλώνα. Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μπορεί να υποφελείται από το ταμείο αυτό, προκειμένου πραγματικά να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία θέλουμε να κατοχυρώσουμε μέσω του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τα οποία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νομικές, νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις για τα κοινωνικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους του κοινωνικού πυλώνα, να έχουμε σημαντικούς επενδικούς στόχους, οι οποίοι να έχουν να κάνουν με τις τομείς του κοινωνικού πυλώνα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, κάτι το, το, το οποίο είπαν οι συνάδελφοι. Η αρχή τη εταιρική σχέση. Συμφωνούμε, η κοινωνία των πολιτών και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι δικαιούχοι. Θα έλεγα και κάτι παραπάνω. Είναι, αν θέλετε, οι φορεί εκείνοι που φέρουν στου ώμου του όλο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τίποτα από όλα αυτά που καταφέραμε στο παρελθόν θα το είχαμε καταφέρει αν δεν είχαμε την συμβολή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τη κοινωνία των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εμπλέκονται στην όλη διαδικασία από την αρχική θέσπιση των προγραμμάτων μέχρι τον τελικό έλεγχο και τις τελικές επιθεωρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν με τη δική τους τη βοήθεια να καταφέρουμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους τους εμπλεκόμενους. Και ένα τελευταίο σημείο το οποίο εθίχτηκε ήδη, το ζήτημα της κοινωνικής ενσωμάτωσης των πιο αποκλεισμένων, των απόρων. Ξέρετε ότι στο παρελθόν, στην προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο, είχαμε το Ταμείο ΦΙΕΤ, το οποίο συνέβαλε και αυτό πάρα πολύ. Αν θέλουμε πραγματικά το 4% στη χρηματοδότηση να γίνει πραγματικός ενωσιακός στόχος, τότε θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο στόχος αυτός χρηματοδότησης για όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον ένα 4% επενδύσει στην κοινωνική ενσωμάτωση. Είδαμε στο παρελθόν ότι χρειαζόμαστε τα χρήματα αυτά. Σαφώ θα πρέπει να γίνει υπό συγκεκριμένων Δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την ε, επιστημιστική βοήθεια, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια περαιτέρω παροχή συμβουλών και πληροφοριών στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση όμω θα πρέπει να έχουμε την επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να έχουμε προγράμματα κοινωνική ενσωμάτωσης να ευχαριστήσω επίσης και την εισηγήτρια για την επέκταση τη ε, καταληκτική ημερομηνία υποβολή τροπολογιών. Σαφώ θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, αλλά και αυτό το λέω προ όλου του συναδέλφου και εκείνου που δεν είναι σκιώδει ηγητέ, είναι εξίσου σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε την ε, οπτική γωνία και αν θέλετε τη συμβολή όλων αυτών των ανθρώπων που συνεργάστηκαν στο παρελθόν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστεί η φωνή του στα πλαίσια τη θέσπιση τη επόμενη ε, χρηματοδοτική περίοδου. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να αφιερώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να ακούσουμε του εμπλεκόμενου φορεί σε όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταλήξουμε στα θετικά αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε από αυτό το Ταμείο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Πρόεδρος χρειάστηκε να φύγει και από ό,τι φαίνεται πρέπει εγώ λέει να την αντικαταστήσω. Ε, που είναι λίγο άβολο τώρα που είμαι και συγκήτρια. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι α, θέλει το λόγο Τόμας Μαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύρια Προεδρεύουσα, αγαπητή Βερόνικα. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή βάση τώρα για την έκθεση αυτή, γιατί εσύ ε, έγραψες την έκθεση. Πάντα οι εκθέσεις σου είναι πάρα πολύ φιλόδοξες, αλλά είσαι προσανατολισμένη και στη συνένεση και έχεις επικοδομητικό πνεύμα και τελικά καταλήγουμε σε καλά αποτελέσματα. Και συμφωνούν όχι μόνο οι Σκιώδης αυτό, αλλά και όλοι μας. Και εγώ τουλάχιστον. Δεύτερον, όταν μας έκανε τις προτάσεις ο Γκιούντερ Ρέτιγκερ, ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό, χάρηκα πολύ γιατί μίλησε για κάποια κέντρα βάρους που θα πρέπει να υλοποιήσουμε. Μεταξύ αυτών είναι το Erasmus Plus. Το Erasmus είναι μια ε, ευρωπαϊκή μάρκα, ένα σήμα εμπορικό ευρωπαϊκό επιτυχίας και υπάρχει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και ε, ε, σε αυτή τη συγκέντρωση στο Erasmus Plus έχει στόχο να αναπτυχθεί το πρόγραμμα. Κάποιοι που γκρινιάζουν ε, ότι χρειάζομαστε περισσότερα λεφτά ή θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δίνουν περισσότερα ή να δούμε ότι αν δεν έχουμε τα χρήματα πώς θα μειώσουμε τις δαπάνες, δηλαδή τα καθήκοντά μας. Όχι, εγώ είμαι υπέρ του πρώτου, να καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι είναι σημαντική η ευρωπαϊκή προϊστηθέμενη αξία και όχι οι εθνικοί εγωισμοί που δυστυχώς τώρα έχουν επικρατήσει και δημιουργούν σχολή. Στην εγγύηση για την νεολαία ισχύει αυτό επίσης. Η εγγύηση για την νεολαία ήταν παιδί του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα κράτη-μέλη αντέδρασαν γιατί ε, οι διοικησει ε, δεν συμφώνησαν, δεν βοήθησαν. Μα όταν έχουμε ε, πρωτοβουλίε για την νεολαία δεν μπορεί να αντιδρούν οι κρατικές μηχανές. Ευτυχώς ασκήθηκε ποιήση και θα πρέπει αυτή να διατηρηθεί και έχει πολύ μεγάλη σχέση και με το Erasmus Plus. Και θα πρέπει όλα αυτά να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Το θέμα είναι να βοηθάμε τους νέους που πρέπει να κάνουν ακροβατικά για να βγουν από την ανεργία. Απίστευτα. Και δεν είναι, ε, βοηθάνε εδώ κούφια λόγια και ανόητα κηρύγματα κυριακάτικα. Ακριβώς θα πρέπει να διατηρηθεί η πίεση για να έχουμε σωστή βάση να προχωρήσουμε. Είδα και τον πρώην Επίτροπο Άντορ. Χαίρομαι που είναι παρόν εδώ. Μεγάλη χαρά. Θυμάται ε, τι έχει γίνει στο παρελθόν και πόσο είχαμε πιέσει, θα διατηρηθεί αυτή η πίεση. Κάτι άλλο, Βερόνικα, είπε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με διάφορα κριτήρια ε, με διάφορους τομείς ε, και θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινωνικά, με τα οικονομικά αλλά και με τα περιφερειακά και τα εδαφικά. Συμφωνώ με τη συνάδελφο Τρεμπέζιος. Δεν πάει να είναι μια χώρα πλούσια. Υπάρχουν πλούσιες χώρες που έχουν φτωχέ περιφέρειες, δυσκολίες προσαρμογής και δεν θα πρέπει να τους κόβουμε τα κονδύλια. Ούτε να έχουμε αυτοματισμούς της μιας περιφέρειας ανάντια στην άλλη. Να έχουν ε, οι άνθρωποι εκεί που το έχουν ανάγκη δυνατότητα να βοηθηθούν. Και τέλος φυσικά οι κοινωνικοί εταίροι να συμμετέχουν ναι με τις συστάσεις αναχώρα, αλλά αγαπητή κυρία Τσίμερ, είναι δύσκολο να φτάνουμε μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού θέλουμε να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Όταν το κάνουμε αναχώρα με ε, ειδικά κριτήρια, ε, είναι καλό αυτό, συμπέρασμα. Νομίζω είναι πολύ καλή βάση για να συζητήσουμε, για να εργαστούμε και με τη βοήθεια των σκιωδών ε, εισηγητών και ο χρόνος είναι λίγος, ας τον αξιοποιήσουμε και είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε. Και είμαστε γνωστοί για τη συνένεσή μας εδώ στην Επιτροπή μας ε, Κοινωνικών Υποθέσεων, πόσο μάλλον όταν η συγκήτρια είναι η Βερόνικα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, Τόμας. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή δουλειά. Δεν ξέρω αν θέλει να μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και η συγγήτρια. Η έκθεση είναι πολύ επικοδομητική. Σίγουρα ένα πολύ καλό σημείο κίνησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους έχουν παρέμβει, τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, διότι ε, ανάμενα και επιπρόσθετες ε, παρατηρήσεις και προσβλέπουμε ε, στις ε, συζητήσεις που θα ακολουθήσουν αυτής και θα σημειώσουμε βέβαια τα σημεία που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής. Θα επικεντρωθώ σε τρεις τεχνικής φύσεως παρατηρήσεις που προέρχονται από τη δική σας έκθεση, που είναι μια έκθεση που αναφέρεται σε προτεραιότητες κλειδιά στις επενδύσεις ε, για τους νέους και για την αύξηση των επενδύσεων για τον τον... την κοινωνική συμπερίληψη και επίσης ε, αναγνωρίζουμε σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με ε, την αιτιολογική έκθεση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την διασφάλιση της προχρηματοδότησης, κυρίως για τα μέτρα της απασχόλησης των νέων. Από τεχνικής άποψης, η προχρηματοδότηση αναφέρεται στις κοινέ διατάξεις, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και ε, εφαρμόζεται οριζόντια στα διάφορα ταμεία, ε, στα ταμεία συνοχής και διαθροτικά ταμεία. Επίσης, η κατεξαίρεση προχρηματοδότηση του 30% ε, παρήχετο για την, ε, για την απασχόληση των νέων το 2015 ε, ήταν μια άπαξ χορήγηση λόγω των οικονομικών περιστάσεων εκείνης της χρονιάς. Ένα άλλο σημείο που θέλω να διευκρινίσω, τεχνικό σημείο, αφορά την προτινόμενη τροπολογία 15, όπου σημειώνουμε ότι η έκθεση αναφέρεται σε πρόταση αύξησης κατά 2% των επενδύσεων ε, στην ε, κοινωνική συμπερίληψη, 2% για τα πρώην μέτρα ΤΕΒΑ, Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους, ειδικά για τη βασική ηλική βοήθεια, που να είναι ε, συμπληρωτικά στο 25% επενδύσεων για την, τον, την κοινωνική συμπερίληψη. Εμείς βλέπουμε την ε, πρότασή μας να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη. Θυμίζω ότι υπάρχουν δύο ειδών κράτη-μέλη ανάλογα με τα επιχειρησιακά προγράμματα που ε, επιλέγουν ε, το επιχειρησιακό πρόγραμμα 1 για την βασική ηλική βοήθεια και το επιχειρησιακό πρόγραμμα τύπου 2 για τα μέτρα συμπερίληψης και τα τελευταία είναι ε, στο φάσμα του 2%. Αυτό απαντά και σε παρεμβάσεις που έχουν γίνει ε, σήμερα σε αυτή την πολύ συζήτηση. Ένα άλλο σημείο, τεχνικό σημείο, έχει να κάνει με την τροπολογία 17, όπου η έκθεση προτείνει ότι ο ειδικός στόχος 11 θα καθορίζεται από το κεφάλαιο 2. Ο ειδικό στόχος 11 είναι ένας ειδικό στόχος που στοχεύει τις δράσεις ε, για την φτώχεια και την βοήθεια, ε, τη βασική ηλική βοήθεια. Θέλουμε να έχουμε ε, τους κανόνες έτσι όπως καθορίζονται σήμερα πιότερους κανόνες και αυτό θα θέλουμε να διέπεται από το κεφάλαιο 3. Τώρα, το πώς μπορούν να διέπονται από το κεφάλαιο 2 ε, αυτό έχει σημασία ε, με τους ε, ισχυρότερους κανόνες και θα εξαρτηθεί από τις δράσεις και τα μέτρα τα οποία θα θέλουμε να κρατήσουμε όσο το δυνατόν πιο ελαφριά. Τα άλλα θέματα, απλούστευση, εταιρική σχέση και εξάμεινο, απλούστευση γενικά. Έχουμε απλούστευση των κανόνων, στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, σε ό,τι αφορά ε, τον προγραμματισμό, σε ό,τι αφορά την διαχείριση και τον έλεγχο, την υποβολή εκθέσεων, τους δείκτες κλπ. Α, οι δύο κανονισμοί θα πρέπει να ε, αναγνωστούν μαζί. Η εταιρική σχέση είναι κλειδί για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι κλειδί για όλα τα ταμεία ε, με τον επιμερισμό της διαχείρισης, διότι ε, αυτό σημαίνει ότι έχει να κάνει με το πώς οι άνθρωποι, οι κοινότητες ή τα εδάφη εισέρχονται σε εταιρικές σχέσεις και αυτό έχει να κάνει και με την πρόταση του ESF, συν όπως το άρθρο 8 αναφέρεται ε, στην επαρκή στήριση στους εταίρους που περιλαμβάνονται, τους κοινωνικούς εταίρους, ως ε, οι κύριοι πρωταγωνιστές, όχι μόνο δικαιούχοι, αλλά κύριοι πρωταγωνιστές και παίκτες ε, στην υλοποίηση των προγραμμάτων επιτόπου. Και τέλος, ευθυγράμμιση με το εξάμεινο, αναφερόμαστε στη σημασία ε, της εστίασης στον κοινωνικό τομέα. Αυτή ήταν η αρχική πρόθεση της Κομισιόν ε, από δύο οπτικές γωνίες. Η αρχιτεκτονική του ιδίου του κανονισμού αντανακλά ακριβώς ε, τους ειδικού στόχους ως εξειδικευμένοι στόχοι για την υλοποίηση του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αλλά όταν μιλάμε για την ευθυγράμμιση με το εξάμεινο, το ίδιο το εξάμεινο αντανακλά ε, ιδιαίτερα στο τομέα της απασχόλησης και τον ελληνικό τομέα, τις αρχές που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό Πύλωνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Με αυτά τα λόγια, κλείνω με πολλές ευχαριστίες από πλευράς Κομισιόν για ένα πολύ ε, καλό σημείο κίνησης ε, με αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θέλει κανένα συνάδελφο να πει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αλλιώ να κλείσει η συζήτηση. Ω εισηγήτρια, το μόνο που θέλω να πω για να κλείσουμε είναι ότι. Καλά, δεν θα πατήσω στι παρατηρήσει των συναδέλφων και των σκιωδών εισηγητών. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μα είπατε και περιμένω με ανυπομονησία όλες τις τροπολογίες. Γιατί πιστεύω ότι συνεργαζόμενοι όλοι μεταξύ μας θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ όλους. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω ότι μπορεί να κλείσει αυτό το θέμα και να περάσουμε στο επόμενο. Έχουμε την παρουσίαση για στιγμή να το βρω. 25 Α, να πω κάτι άλλο προηγουμένω. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών για την έκθεσή μου 25 Σεπτεμβρίου. Παρατάθηκε λίγο η ε, προθεσμία. Το ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, αλλά αναγκαστήκαμε να το κάνουμε. 18 Οκτωβρίου θα το συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή και θα ψηφίσουμε εν ευθέτω χρόνο 26 και 27 Νοεμβρίου και ελπίζω να προλάβουμε με καλές συμβαστικές προτάσεις να το διεκπαιρεώσουμε στην τελευταία ολομέλεια τον Απρίλιο πριν τις εκλογές. Να εγκριθεί η έκθεση δηλαδή. Αυτά. Y ahora vamos a pasar al segundo Το δεύτερο θέμα για σήμερα είναι το εργαστήριο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus. Θέλω να ευχαριστήσω τους συγητές μας και ιδιαίτερα τον πρώην Επίτροπο και φίλο ε, ε, Άντορ, στον οποίο και δίνω μέσα στο λόγο. Good afternoon, ε, Madam Chair. Καλησπέρα σας, ε, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Η αίθουσα αυτή, η επιτροπή αυτή μου φέρνει στο νου πολύ ευχάριστα αναμνήσεις για μένα. Θα ήθελα να σας πω βέβαια εξ αρχής ότι μιλώ σήμερα εδώ για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τον παλαιό και τον νέο κανονισμό σαν εξάρτητος παρεμβαίνων που έχει βέβαια πολύ καλή μνήμη. Και θα ήθελα να σε υπενθυμίσω κάποια από τα βασικά στοιχεία του προηγούμενου χρηματοδοτικού κύκλου, τα οποία θα πρέπει να συγκρίνουμε με τον επόμενο κύκλο χρηματοδότησης. Στα 10 λεπτά που έχω στη θέση μου, θα ήθελα να τονίσω λίγο πώς έχει εξελιχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο γίνεται πλέον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, Θα θέλαμε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των προγραμμάτων κάθε χώρας και να καταφέρουμε να δούμε επίσης και μια σειρά από προτινόμενες λύσεις. Για να συνδέσω την παρουσίασή μου αυτή με τη συζήτηση που μόλις τώρα έγινε, θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποιες προτάσεις του 2010, όταν η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συζητώντας το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο τότε, είχε κάνει συγκεκριμένε προτάσεις για συγκεκριμένα ποσά. Βλέποντας τα ποσά αυτά συνειδητοποιούμε ότι ε, πάρα πολλέ από τις ιδέες που ακούμε σήμερα είχαν ήδη ακουστεί από τότε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια από τη μία περίοδο προγραμματισμού στην άλλη να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Ταμείου αυτού και να συμπεριλάβουμε νέα καινοτόμα στοιχεία όσον αφορά νέες προϋποθέσεις, όσον αφορά τους νέους κανονισμούς, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε πιο θετικά αποτελέσματα. Ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα μια εξέλιξη, αν θέλετε, του Ταμείου και όχι μια επαναστατική αναμόρφωσή του. Σας καλώ τώρα να συγκρίνουμε λίγο τις προσπάθειες που γίνανε από την Επιτροπή Μπαρόζο σε σχέση με αυτές που γίνανε από την Επιτροπή Γιούνκερ σε πέντε συγκεκριμένους τομείς, έξι μάλλον για την ακρίβεια. Να δούμε καταρχάς πώς καθορίζεται το συνολικό ποσό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, πώ πετυχαίνουμε την καλύτερη ευθυγράμμιση πολιτικών, τι γίνεται με την κοινωνική ενσωμάτωση, τι γίνεται με τους νέου, πώ έχουμε καλύτερη χρηματοδότηση και καλύτερη διαβίβαση των πόρων από άλλα ταμεία προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τι μπορούμε και εμείς και εσείς να κάνετε όσον αφορά την απλούστευση. Στον προηγούμενο κύκλο προγραμματισμού, που ουσιαστικά είναι η τρέχουσα πλέον περίοδο για το πολιτέ νομοσυνομικό πλαίσιο, έχουμε ένα καινοτόμο στοιχείο προκειμένου να θεσπίσουμε καλύτερα το συνολικό ποσό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα πλαίσια του κοινωνικού προϋπολογισμού. Ξέρετε ότι για ένα ταμείο το οποίο εντάσσεται στο Ταμείο Συνοχής υπήρχε μια κάποια αυτονομία από τα κράτη-μέλη. Καταβλήθηκε λοιπόν μια μάχη θα έλεγα ακόμα για να καταφέρουμε να θεσπίσουμε καλύτερα το συνολικό ποσό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ως ποσοστό πλέον του Ταμείου Συνοχής. Και αυτό εξελίχθηκε πλέον σε ένα τελικό ποσό, σε ένα απόλυτο ποσό, το οποίο ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για την εφταετή αυτή περίοδο από το 2021 στο 2027. Πρέπει να δούμε πώς αυτά τα 101,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα χρησιμοποιηθούν στην πράξη. Το μήνυμα πάντως είναι ξεκάθαρο. Δεν μιλάμε πλέον για ένα απόθεμα, για κάτι το οποίο περισσεύει από άλλα ταμεία, αλλά κάτι το οποίο θεσπίζεται εξ αρχής και χρησιμοποιείται στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού. Όσον αφορά τώρα την ευθυγράμμιση πολιτικών, στον προηγούμενο κύκλο προγραμματισμού μέχρι το 2020 δηλαδή, που θα έπρεπε να εφαρμοστεί μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Έχουμε νέα καινοτόμα στοιχεία, όπως τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αναφέρθηκαν σε αυτό πολλοί ομιλητέ και έχουμε πλέον μια πιο στενή διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε περισσότερο την κατεύθυνση αυτή όσον αφορά την αρμόνιση και την ευθυγράμμιση των πολιτικών. Τώρα, κοινωνική ενσωμάτωση. Θα περάσουμε από το 20% στο 25%. Αναφέρθηκαν σε αυτό πολλοί ομιλητέ. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω στο σημείο αυτό και για λόγου, αν θέλετε ιστορική αναδρομή, δεν θα πρέπει να θεωρήσετε ότι αυτό το 20% είναι απόλυτα διαθέσιμο και μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε, ότι είναι απόλυτα δεδομένο. Όταν προτάθηκε αυτό το 2011, δεν μπορώ να σας πω πόσοι πολλοί άνθρωποι μου είπαν τότε ότι ήταν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο και το Συμβούλιο θα πέριπτε την πρόταση αυτή. Και υπήρχε και μια άλλη επιτροπή του Κοινοβουλίου αυτού που θα πέριπτε αυτή την πρόταση, όχι προφανώ η δικιά σα. Και ότι θα υπήρχαν και πολλέ ομάδε ενδιαφερομένων μερών που ουσιαστικά θα πέριπταν αυτό το προτινόμενο ποσοστό. Τελικά διατηρήθηκε το 20% θεσμοθετήθηκε, μολονότι χρειάστηκε να υπερκεράσουμε πολλές δυσκολίες. Και ο τότε, πρόεδρο, και ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόσο, είχε κάποιους ενδιασμούς για το θα έπρεπε να διατηρήσουμε το ποσοστό αυτό. Και πραγματικά θα μπορούσα να σας πω πως πριν από 7 χρόνια κατάφερα τελικά με πολλές προσπάθειες να πείσω τον πρόεδρο Μπαρόσο να διατηρήσει το 20% για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όχι μόνο να δούμε ότι παραμένει το ποσοστό αυτό, αλλά ότι προτείνεται και αύξησή του στο 25%. Όσον αφορά τώρα την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ενσωματώνεται και αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υπάρχει, αν θέλετε, ο δικό τη χρηματοδοτικό ε, φάκελο. Στον ε, πίνακα αυτό συγκρίνουμε πώς έχουν τα πράγματα με την υφιστάμενη περίοδο σε σχέση με αυτά τα οποία προτείνονται για την ε, επερχόμενη περίοδο προγραμματισμού. Αν δούμε τι προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011, στην ε, απαρχή δηλαδή των διαπραγματεύσεων όσον αφορά την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, η απάντηση είναι τίποτα απολύτω τότε. Και αυτό διότι θεωρούσαμε ότι οτιδήποτε μπορούσε να χρηματοδοτήσει το ταμείο αυτό θα μπορούσε τελικά να επιτευχθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αποφασίσαμε τελικά όμω να ενσωματώσουμε την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων προκειμένου να προβληθεί περισσότερο και προκειμένου να μπορούν και οι εθνικές αρχέ να επιβλέπουν περισσότερο την εφαρμογή μια πολιτική που είχε τότε πάρει και το πράσινο φω από το Συμβούλιο και αναφέρομαι βέβαια στην εγγύηση για την νεολαία. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να κρατήσουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και το πρόγραμμα αυτό με τον ξεχωριστό προπολογισμό, ο οποίο έχει επιβεβαιωθεί. Όσον αφορά τώρα την ε, δυνατότητες διαβίβασης των χρηματοοικονομικών πόρων, αυτό το οποίο βλέπετε με τον όρο engineering στην διαφάνεια. Εδώ πέρα πάλι θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στα όσα προβλέπονται. Στον προηγούμενο κύκλο προγραμματισμού και χρηματοδότησης είχαμε δημιουργήσει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποια επιπλέον ποσά, επιπλέον πόρους για τοπικές κυβερνήσεις προκειμένου να προωθήσουν κοινωνικές πολιτικές. Παρ' όλα αυτά παραδέχομαι ότι οι πρωτοβουλίες αυτές είναι αρκετά περιορισμένες. Η πρόθεση λοιπόν τώρα είναι να καταφέρουμε να έχουμε περισσότερε επενδύσει και μια ισχυρότερη χρηματοδότηση με θετικέ κοινωνικέ συνέπειε. Σαφώ λοιπόν η συμπερίληψη των νέων αυτών πόρων είναι σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κοινωνική καινοτομία, αλλά θα πρέπει επίση να δούμε και πού πραγματικά εστιαζόμαστε, που εστιάζεται το Ταμείο αυτό και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλίνουμε από τους βασικούς στόχους. Όσον αφορά τον στόχο της απλούστευσης, ξέρετε ότι εδώ πέρα έχουμε τις, τα καταποκοπήν ποσά, καθώς επίσης και τις ε, επιλογές απλούστευσης του κόστους, αυτή τη στιγμή ε, ενσωματώνονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Πλάς και άλλα επιμέρους μικρότερα ταμεία, μας δίδεται κατάλληλη ευκαιρία για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή απλούστευση. Πάντα βέβαια υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τελικά καλύτερα και την ευθυγράμμιση των πολιτικών των κρατών μελών και θα διασφαλίσει εν τέλει ότι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα θα μπορούν να εφαρμοστούν και στην πράξη. Τώρα πολύ συχνά αξιολογούμε τις επιδόσεις των κρατών μελών και τις επιδόσεις των χρηματοδοτικών αυτών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της απορρόφησης. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα τώρα να επικεντρωθώ, λέγοντας βέβαια ότι αποτελεί μόνο ένα από τα πολλά σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Η απορρόφηση λοιπόν, το ποσοστό απορρόφησης αποτελεί έναν, μια παράμετρο ροής. Ε, είναι μία παράμετρος που λαμβάνεται επίσης υπόψη σε σχέση με άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα όταν τηρούνται όλες τις τυπικές διαδικασίες και προσπαθούμε επίσης σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη να δούμε τελικά αν μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πετυχαίνουμε ή όχι σύγκληση. Στον πίνακα λοιπόν αυτό βλέπετε στην αριστερή πλευρά όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε input, τις ροές, και στη δεξιά πλευρά αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε output. Εξωτερικούς και εσωτερικούς τελικά παράγοντες, ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες που καθορίσουν τελικά την καλή εφαρμογή των προγραμμάτων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να λεφθούν υπόψη σε οποιαδήποτε αξιολόγηση γίνεται. Όσον αφορά του ε, φορεί εφαρμογή τη κοινωνική πολιτική, το πιο σημαντικό είναι να δούμε αν πετυχαίνουμε τελικά κοινωνική σύγκληση. Αν θέλουμε όμω πραγματικά τα ταμεία αυτά να προωθούν τις πολιτικές, τότε η απορρόφηση των πόρων από τα ταμεία αυτά γίνεται πολύ σημαντικό ζήτημα. Αν έχουμε χαμηλό ποσοστό απορρόφησης, αν υπάρχει πολύ μεγάλη διακύμανση στο ποσοστό απορρόφησης, τότε κατά πάσα πιθανότητα η συγκεκριμένη αυτή πολιτική δεν θα εφαρμοστεί σωστά, ούτε θα προχωρήσουμε στον ευκταίο μετασχηματισμού. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί παράγοντες, πολιτικοί, οικονομικοί και διοικητικοί λόγοι που δικαιολογούν αυτή τη χαμηλή απορρόφηση. Διοικητικέ δυναμίε, για παράδειγμα, μπορεί να εξηγήσουν μια τέτοια χαμηλή επίδοση, οι επιδόσεις παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσει. Ας μην σα τρομάξουν στη διαφάνεια αυτή όλα αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, τα οποία ουσιαστικά σα περιγράφουν συνοπτικά την όλη εμπειρία την οποία έχουμε συσσωρεύσει από τον προηγούμενο κύκλο χρηματοδότηση και προγραμματισμού. Βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχουν χώρε οι οποίε καταφέρνουν σε μια περίοδο προγραμματισμού να απορροφήσουν πολλέ φορέ ακόμα και το 90% των διατηθέμενων πόρων, ενώ άλλε χώρε κυμαίνονται στο 50, 60, 70%. Μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερα προβληματικές περιπτώσεις και βάσει των αριθμητικών αυτών δεδομένων που είδατε στην προηγούμενη διαφάνεια, μολονότι ήταν βέβαια τα γράμματα πολύ μικρά για να τους διαβάσετε, μπορούμε εδώ πέρα να καταλήξουμε στις διαφορετικές κατηγορίες. Έχουμε ουσιαστικά χώρες με ισχυρές ή αδύναμες διοικητικές ε, δομές, οι χώρες οι οποίες έχουν χαμηλό ή υψηλό ποσοστό ευθυγράμμιση όσον αφορά την πολιτική. Και από κοινού τα στοιχεία αυτά τελικά καθορίζουν το αν μια χώρα είναι σε θέση να απορροφήσει ή όχι τους απαραίτητους πόρους. Βλέπετε ότι η Αυστρία αποτελεί μια χώρα πρωταθλητή, έχει καταφέρει τελικά να απορροφήσει του πόρου πόρους προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 90%. Η Ισπανία κατάφερε να εντοπίσει τι κατάλληλε πολιτικέ, αλλά οι εθνικέ τη δομέ είναι αρκετά πολύπλοκε. Οι εθνικέ εγχώριε δομέ της Ισπανία ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκε για να επιτρέψουν καλύτερη απορρόφηση των πόρων, με αποτέλεσμα τελικά το ποσοστό απορρόφησης Ισπανίας να είναι πολύ χαμηλό. Έχουμε την, το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει πολύ χαμηλό ποσοστό σφάλματο, πολύ καλέ διοικητικέ δομέ αλλά δεν έχει καταφέρει να εγκρίνει προγράμματα τα οποία να συνάδουν με τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική πολιτική. Γι' αυτό το λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ποσοστό απορρόφησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι χαμηλό. Η Ρουμανία από την άλλη έχει και αδύναμες διοικητικέ δομές και ένα χαμηλό ποσοστό ευθυγράμμιση όσον αφορά τον τομέα πολιτικής. Αν δούμε για παράδειγμα την ενσωμάτωση των Ρωμάν στην κοινωνία ή την καλύτερη ενσωμάτωση της, των Ρωμά στην αγορά εργασία, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ πέρα οι επιδόσεις της Ρουμανίας ήταν πολύ χαμηλές. Και γι' αυτό το λόγο τελικά και η απορρόφηση των πόρων ήταν και αυτή ιδιαίτερα χαμηλή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε τις κατηγορίες αυτές ξεχωριστά και από κοινού και θα πρέπει έπειτα όταν ψάξουμε να δούμε τελικά πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να δούμε και ποιοι είναι οι τελικοί αποδέκτες των πόρων αυτών, τι γίνεται δηλαδή σε εθνικό επίπεδο και α μην ψάξουμε του υπέτειου μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για χαμηλή απορρόφηση πόρων από άλλα ταμεία, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Και εκεί πολλέ φορές έχουμε χαμηλή απορρόφηση των πόρων με αποτέλεσμα τελικά να παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο η ίδια διαβίβαση των πόρων στους τελικούς αποδέκτες. Και σε ορισμένε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε ακόμα και αντίδραση στη χρήση ή απόρριψη της χρήσης του ταμείου αυτού. Και μάλιστα Ξέρετε ότι ε, αν είχε χρησιμοποιηθεί το ταμείο αυτό εκτενέστερα στην Ευρωπαϊκή, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να σας πω ότι και η άποψη πολλών Βρετανών, ιδίω στη Βόρεια Αγγλία που πλήττεται από ανεργία, θα ήταν εντελώ διαφορετική όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είχαν αποφεληθεί πραγματικά από τους πόρους του ταμείου αυτού. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα τη προχρηματοδότηση. Εδώ πέρα είχαμε εντοπίσει κάποια προβλήματα στο παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο η τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάποιε αλλαγέ στην προχρηματοδότηση. Α μην ξεχνάμε εδώ πέρα τι δυνατότητε προχρηματοδότηση στα πλαίσια τη πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ε, ένα σκέλο το οποίο θα πρέπει να διατηρηθεί και μετά την ενσωμάτωση πρωτοβουλία αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο όσον αφορά την μικροχρηματοδότηση. Και εδώ είχαμε κάποια προβληματικά σημεία. Χρειάστηκε εδώ πέρα να καταφέρουμε να συνεργαστούμε περισσότερο με το EIF και να καταφέρουμε εδώ πέρα να επιλύσουμε τα προβλήματα τα οποία είχαν ε, εντοπιστεί στο παρελθόν. Θα πρέπει τώρα να προχωρήσω γρήγορα. Τώρα, πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα απορρόφησης. Ας ξεκινήσουμε από τις λύσεις που εντοπίσαμε και στο παρελθόν. Ευελιξία, απλούστευση. Αυτέ, αν θέλετε είναι οι πιο τυποποιημένε λύσει, αλλά δεν λύνουν πλήρως το πρόβλημα. Η απλούστευση είναι, αν θέλετε, μία λύση ιδιαίτερα ελκυστική. Δίνουμε τη δυνατότητα πρόσβαση σε περισσότερους πελάτες εντό αγωγικών, σε περισσότερους αποδέκτες, μεγαλύτερη ευελιξία. Μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε τι απαραίτητε προσαρμογές και αλλαγέ. Το πρόβλημα όμω είναι ότι η απλούστευση πολλέ φορέ απορρέει από το εθνικό επίπεδο, ενώ οι αλλαγέ οι οποίε προτείνονται και επιβάλλονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να μην επιφέρουν τελικά λύσει. Η ευελιξία από την άλλη, αν είναι υπερβάλλουσα, τότε πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε ένα ESF, στην Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο θα εξυπηρετεί με μονομένε ανάγκε και δεν θα λειτουργήσει λογικά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ πέρα να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία, να αποφύγουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν λόγω παρατυπιών. Και α μην ξεχνάμε εδώ πέρα ότι πολλέ φορέ η υπερβολική ευελιξία μπορεί να μα εμποδίσει να ευθυγραμμιστούμε με τι κεντρικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντα όλα αυτά κατά νου, θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μία άλλη κατεύθυνση. Να δυναμώσουμε περισσότερο του τοπικού παράγοντε. Δεν σημαίνει αυτό ότι δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Σημαίνει ουσιαστικά ότι δίνουμε μεγαλύτερη δύναμη, περισσότερε αρμοδιότητε στο τοπικό επίπεδο για να συνδεθεί καλύτερα με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Να σα δώσω τρία παραδείγματα. Ενσωμάτωση των μεταναστών. Σίγουρα εδώ πέρα δεν μπορούμε να βρούμε μια μαγική λύση για όλου. Ενδεχομένω οι πόλει σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο πόλων να γνωρίσουμε καλύτερα τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε με τους μετανάστες. Και ίσως θα πρέπει ακριβώς οι πόλεις αυτές να μπορούν να κάνουν άμεσα αιτήσει. Κοινωνική εταίρεια συνεχεία. Δυστυχώς πολλές φορές η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων επηρεάζεται από ε, πολιτικά συμφέροντα σε τοπικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν και οι κοινωνικοί εταίροι να ξεφεύγουν, αν θέλετε, από του περιορισμού που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο και να υποβάλουν αιτήσει άμεσα. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το EGF, αναφέρθηκα στο Ηνωμένο Βασίλειο και η δική μου χώρα, η Ουγγαρία, πολλέ φορέ δεν προστρέχει στο ταμείο αυτό. Θεωρώ ότι πάλι εδώ πέρα οι περιφέρειε σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2 έχουν πολύ περισσότερε γνώσει και είναι σε θέση να ξέρουν αν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το EGF ή όχι. δίνω κάποια κάποια ενδεικτικά παραδείγματα δεν θεωρώ ότι εδώ πέρα θα πρέπει να βρεθεί κάποια επαναστατική λύση. Νομίζω θα πρέπει να διευθετήσουμε καλύτερα, να προσαρμόσουμε καλύτερα τα εφιστάμενα εργαλεία και μέσα που έχουμε για να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αν πιάνει τα πέντε συμπεράσματα στα οποία καταλήγω στην παρουσίασή μου αυτή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εστιαστούμε στον στόχο των ταμείων αυτών, είτε πρόκειται για το σύνολο του κοινοτικού προπολογισμού, είτε πρόκειται για επιμέρου εργαλεία ή προγράμματα. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην διοικητική ικανότητα των κρατών μελών με τους απαραίτητους περιορισμούς όμως, γιατί η διοικητική ικανότητα δεν είναι το μόνο ζήτημα, θα πρέπει να διευθετηθούν και άλλα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να καταφέρουμε να έχουμε καλύτερο ανιστερνισμό των προγραμμάτων αυτών, καλύτερη εμπλοκή του τοπικού επίπεδου, αύξηση της συμμετοχής αύξηση του ποσοστού της χρηματοδότησης και να μπορούμε να έχουμε μία διαχείριση η οποία δεν θα είναι μόνο άμεση και έμεση, αλλά θα δίνει μεγαλύτερο βάρος και στην επιμερισμένη πτυχή, στην επιμερισμένη διαχείριση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Άντορ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όσο και εξαντλητική η παρουσίασή σας. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Σάμεκ, που είναι η πρόεδρος ε, και αρμόδια για να μιλήσει για αυτά τα θέματα για την τρέχουσα περίοδο. Έλεγα ότι είναι η πρόεδρος και διευθύντρια του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας από την Ιταλία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την συνάντηση. Αυτό ήταν ένα σημείο ανημέρωση που είχαμε ετοιμάσει για αυτή την Επιτροπή στην αρχή του χρόνου, δηλαδή πριν από τις νέες προτάσεις για τον ε, κανονισμό ESF+. Και είχαμε εστιάσει την προσοχή μας κυρίως στο πώς θέλουμε να επεκτείνουμε τις κανονιστικές αλλαγές ε, που έχουν εισαχθεί και πώς έχουν επηρεάσει την υλοποίηση των προγραμμάτων. Και βλέπουμε τώρα, ε, εστιαζόμαστε κυρίως στην απλούστευση και την διοικητική ικανότητα. Κάναμε μια αναθεώρηση των εγγράφων επί χάρτου, αλλά κάναμε και κάποια δουλειά επί τόπου. Ε, Διεξαγάμε συνεντεύξεις, έρευνες, ε, επικοινωνήσαμε με 90 ε, περίπου συμμετόχους, ενδιαφερομένα μέρη, δικαιούχους, διαχειριστικές αρχές και εμπειρογνώμονες. Τώρα, ποια είναι τα κυριότερα θέματα που έχουν προκύψει σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που προέκυψαν σε αυτή την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. ποιε είναι αυτές που θεωρούνται πιο συναφείς από τους δικαιούχου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Η πρώτη ήταν η ισχυρότερη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην αύξηση χωρίς αποκλεισμού. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η συγκέντρωση στην κοινωνική ένταξη, το 20% το πόσο στο που θα δαπανηθεί σε αυτό το μέτρο σημαίνει ότι ε, συμμετείχαν νέοι δικαιούχοι σε αυτό το ταμείο, νέες δράσεις προωθήθηκαν που αυτό διαφέρει από τις συνήθεις της προηγούμενες ε, δράσεις και μέτρα του ΕΚΤ, όχι μόνο εκπαίδευση, αλλά πιο ε, πολλά μέτρα κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης. Και επίσης νέοι συμμετέχοντες, νέες ομάδες στόχου, όχι μόνο οι άνεργοι, αλλά και πολλές μειονιστούσες ομάδες, ε, οι Ρωμά, οι μετανάστες, ε, οι άστεγοι κλπ. Και όπως είπα, έχουμε νέους δικαιούχους. Δηλαδή, δεν έχουμε τους συνήθεις υπόπτους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, αλλά και κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δήμοι κλπ που ε, διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο όπως έχει ήδη Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε κατά νου, διότι αυτό επηρεάζει την αντίληψη αυτών των δικαιούχων για τις αλλαγές, για τα κυριότερα θέματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη νέα προγραμματική περίοδο. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές αλλαγές είναι αυτή η αναγνώριση ότι το σύστημα υλοποίησης απλουστεύτηκε σε σχέση με προηγούμενες περιόδους προγραμματισμού, αλλά για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν είναι και τόσο μεγάλη αλλαγή, γιατί και στην προηγούμενη περίοδο του 7 έως 13 το ESF ήδη είχε δοκιμάσει να απλουστεύσει ε, το σύστημα υλοποίησης ε, και το ε, σύστημα των απλουστευμένων επιλογών κόστους. Και ήταν δυνατόν επίσης και με τον κανονισμό ΕΚΤ να δοθεί δυνατότητα στην Κομισιόν να υιοθετήσει νέες απλουστευμένες επιλογές ε, κόστους με κατεξουσιοδότηση πράξης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους δικαιούχους και τις διαχειριστικές αρχές, διότι εκεί υπήρχε μεγαλύτερη ασφαλεία δικαίου σε αυτού του τύπου τις επιλογές που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Και επίσης κάτι άλλο, αυτό συνεπάγεται χαμηλότερο ε, ποσοστό σφάλματος και χαμηλότερο διοικητικό φόρτο και για τις διαχειριστικές αρχές και για τους δικαιούχους. Τα άλλα δύο σημαντικά θέματα τα οποία υπογραμμίστηκαν από τους ίδιους τους δικαιούχους ήταν οι διατάξεις δημιουργίας ικανοτήτων, ειδικέ διατάξεις που ζητούν ζητάνε από τη διαχειριστική αρχή να διευκρινίσει τις δράσεις δημιουργίας ικανοτήτων που θα υλοποιήσουν και ε, σε επιχειρησιακά προγράμματα και σε εταιρικές σχέσεις. Και επίσης υπάρχει επικέντρωση στην συνεργασία, στην εταιρική σχέση. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα, πιο σημαντικές ε, αλλαγές ε, τις οποίες ε, έχουν υποδείξει ήδη οι δικαιούχοι. Και από τις συνεντεύξεις έχουμε επιβεβαιώσει αυτό που έχουμε δει και σε μελέτες που έχουν ε, διεξαχθεί πρόσφατα τα πρόσφατα χρόνια ε, για λογαριασμό της Κομισιόν. Ποιοι είναι οι κυριότεροι τομείς προβλημάτων, ιδιαίτερα για τους νέους δικαιούχους, όπως είπα, η ΜΚΟ, Δήμοι, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κυρίως για μικρούς δικαιούχους, που είναι κυρίως αυτοί που έχουν τις πιο καινοτόμες ιδέες για το πώς να επιλύσουν προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, αλλά δεν ε, γνωρίζουν τους κανόνες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και τους ε, ε, βρίσκουν πολύ δύσκολους στην εφαρμογή. Ε, στον κύκλο του, των προγραμμάτων. Στην αρχή υπάρχουν ε, προβλήματα. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση, στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Λένε οι δικαιούχοι ότι υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας για ευκαιρίες. Δεν γνωρίζουν πότε υπάρχουν αυτές οι ε, ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του ΕΚΤ και δεν υπάρχει βοήθεια αν θέλουν να υποβάλουν μια αίτηση ε, σε κάποια πρόσκληση υποβολής ε, προτάσεων, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουν σε ποιον αποταθούν, με τις απορίες τους, ποιος μπορεί να τους βοηθήσει στην προετοιμασία των προτάσεών τους. Και αυτό γιατί υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες από ταμείο σε ταμείο και από διαχειριστική αρχή σε διαχειριστική αρχή. Ακόμη και στην ίδια περιφέρεια, στο ίδιο πρόγραμμα, μερικές φορές, για παράδειγμα, κοινωνική ένταξη. Ε, αυτός ο άξονας ε, εμπίπτει σε διάφορους φορείς, ανάλογα ε, με αν είναι απασχόληση ή εκπαίδευση. Και πολύ συχνά είναι δύσκολο να ε, κατανοήσουν τους ε, επιμερούς κανόνες. Ε, υπάρχουν προθεσμίες, πολύ στενές προθεσμίες. Συνήθως είναι δύο μήνες. Είναι πολύ μικροχρονικό διάστημα, ιδιαίτερα αν θέλει κανείς να προτείνει ε, κάτι νέο, ένα περίπλοκο, μια καινοτομία. Και είναι πολύ μικρή προθεσμία για να δημιουργηθούν αποτελεσματικές εταιρικές σχέσεις. Επίσης, άλλο πρόβλημα, η χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην πραγματικότητα συνήθως ε, θεωρούνται πολύ περιπλοκές και άκαμπτες ε, γιατί σχεδιάζονται με βάση τις συνήθεις ε, δραστηριότητες του ESF, εκπαίδευση, κατάρτιση και είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν για άλλου τύπου προγράμματα. Άλλο πρόβλημα ε, η διαδικασία είναι μακράς διάρκειας, δεν είναι διαφανής διαδικασία επιλογής και σε πολλές χώρες είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποιος είχε επιλεγεί, ποια έργα έχουν επιλεγεί και για ποιους λόγους έχουν γίνει αυτές οι επιλογές. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, την υλοποίηση των έργων και πάλι ε, από αυτά που μας είπαν οι δικαιούχοι. Υπάρχουν υπερβολικά πολύ περίπλοκοι κανόνες επιλεξιμότητας, ε, τεκμηρίωση και έγγραφα που πρέπει να συλλεγούν ε, και αιτιολογικά. Ε, υπάρχουν επικαλύψεις κανόνων, ευρωπαϊκοί κανόνες, εθνικοί, τοπικοί, περιφερειακοί κανόνες ε, όταν τα προγράμματα τη χάνουν διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο. Πολλαπλά αντικείμενα αναφορά με διαφορετικέ ερμηνείε, ε, κανόνε επιλεξιμότητε, ιδιαίτερα για μικρού δικαιούχου. Ένα πρόβλημα είναι ότι έχουν περιορισμένη διοικητική και διαχειριστική ικανότητα. Πρέπει να μάθουν πώς να διαχειρίζουν αυτού του τύπου τα προγράμματα. Και τέλος, η επιλεξιμότητα τα ε, δαπανών και η απέτηση υποβολής εκθέσεων. Ε, υπάρχει ε, τεράστιο χαρτοβασίλειο, υπάρχει διαδικασία ελέγχων επιθεωρήσεων σε, επιθεωρήσεων σε πολλαπλά επίπεδα. Πολλές φορές τη χάνουν διαφορετικής ερμηνείας, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια σε ό,τι αφορά το τύπο του, της δαπάνης που θα καλυφθεί, ε, υπερβολική συλλογή δεδομένων, αναφορές, αρχαιοθέτηση και καθυστερημένες πληρωμές. Κάποιοι δικαιούχοι μας είπαν ότι καθυστερούν πληρωμές ακόμη και 12-18 ε, μήνες μετά. Εδώ έχουμε κάποιους αριθμούς με τα αποτελέσματα των ερευνών μας που δείχνουν με πράσινο βλέπουμε τους δικαιούχους που λένε ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, οι ενάγκες τους έχουν ε, αντιμετωπιστεί, με το κόκκινο δεν έχουν αντιμετωπιστεί, βλέπουμε ότι πολλά πράγματα δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Ιδιαίτερα το χάσμα σε ό,τι αφορά τους κανόνες και τους κανονισμούς, τους ελέγχους και τις ε, επιθεωρήσεις, ε, ότι τα συστήματα δεν λειτουργούν καλά, τα, τα, συστήματα πληροφορικής. Τώρα, η χρήση και η χρησιμότητα των εργαλείων, οι περισσότεροι δικαιούχοι μας είπαν ότι τα πιο σημαντικά ήταν η κατηξουσιοδότηση ε, πράξης ε, για ε, τις απλουσευμένες επιλογές κόστους. Τα κράτη-μέλη έχουν εισάγει κάποια μέτρα για να στηρίξουν τους δικαιούχους, αλλά αυτά δεν ήταν επαρκή. Σύμφωνα με τους περισσότερους δικαιούχους που έχουμε, στους οποίους έχουμε απευθυνθεί και στο τέλος αυτό που λένε οι δικαιούχοι είναι ότι το διοικητικό φορ, ο διοικητικός φόρτος είναι ε, θέμα, είναι ένα πρόβλημα για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, το πρόβλημα του πώς ε, να κάνουν ε, το πρόγραμμα του ESF να μπορεί να συμπεριλάβει καινοτόμα έργα και να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις. Και το άλλο ήταν ο κίνδυνος περικοπών του προπολογισμού. Σε ό,τι φορά τις συστάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε τις απλουστευμένες δομές, λιγότερες, πιο σαφή, λιγότερο πιο σαφείς ε, ε, κανόνες, εκτεταμένη χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών και επιλογών κόστους. Το θέμα εδώ είναι να είμαστε προσεκτικοί όμως σε ό,τι αφορά τις απλουστευμένες επιλογές κόστους, να, να προσοχή για το ε, συγκεκριμένο περιεχόμενο των, της δράσης ESF, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στην κοινωνική ένταξη. Γιατί όταν μιλάμε για τα αποτελέσματα, και την αποδοχή των δαπανών σύμφωνα με το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να θεωρούμε μόνο την κατάσταση απασχόλησης ένα, καλό αποτέλεσμα, διότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι ένας καλός ε, δείκτης. Ένα μεγάλο ε, πρόβλημα είναι η ικανότητα ε, υποδομών. Η, θα πρέπει να υπάρχουν δράσεις ε, δυνατότητας δημιουργίας ε, υποδομών και ικανοτήτων. Ιδιαίτερα με το esf sin που, όπου συγχωνεύονται διαφορετικά ταμεία, όπου θα υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις ε, και γνώσεις που θα συγχωνευτούν για παράδειγμα με τον επιμερισμό των πρακτικών και της δράσης αμοιβαίας γνώσης, ε, μάθησης και ένα άλλο σημαντικό θέμα, η ισχυρότερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και όχι μόνο των κοινωνικών εταίρων, αλλά και των δήμων, των πόλεων, των κοινοτήτων, των ε, ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, διότι είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό των απλουστευμένων μεθόδων που θα μπορούν να προωθήσουν ε, πετυχεμένες δράσεις και θα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στο να δημιουργήσουν οδηγίες, κατευθυντήρες γραμμές και οδηγούς που είναι ε, χρήσιμοι για την ομαλή συνέχιση του προγράμματος. Αυτοί οι νέοι ενδιαφορούμενοι φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν από την αρχή κιόλας ε, του σχεδιασμού του προγράμματος μέχρι την υλοποίηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Σαμέκ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπροζαίτης, ο οποίος είναι διοικητικός διευθυντής του, συστήμα, του Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής και Δημόσιας Διαχείρισης στη Λιθουανία. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα και να ακούσω και από εσά ποια είναι τα διδάγματα, τα συμπεράσματα των μελετών που έχει διεξάγει το Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρώτερη και την υφιστάμενη προγραμματική περίοδο για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και πώς μπορεί αυτό να επιτευχθεί περισσότερο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. και όλους ιδιαίτερως βέβαια μέσω του ΦΕΑ, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους άπορους. Θα ήθελα στο λίγο χρόνο που έχω στη θέση μου να δούμε πολύ γρήγορα μαζί την πολύπλοκη αυτή πρόκληση της παιδικής φτώχειας, πώς αξιολογείται, πώς προσμετάται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούμε να την προσεγγίσουμε ενοιολογικά, ποια πολιτική εγκρίνουν τα κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουν την παιδική φτώχεια, να δούμε τι κάνει το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, όπου εκεί πέρα μπορούμε να δούμε και κάποιες συγκεκριμένες πρακτικές και προτάσεις βελτίωσης για την επερχόμενη περίοδο προγραμματισμού. Η παιδική φτώχεια από μόνη της είναι ένα ζήτημα πολυδιάστατο. Πολλοί θεωρούν ότι η παιδική φτώχεια έχει να κάνει μόνο με την, ηλική, με την φτώχεια, με την έλλειψη χρημάτων. Στην πραγματικότητα είναι μια ένδια που οδηγεί σε μια πολυδιάστατη τελικά φτώχεια που πλήττει τα παιδιά. Αποτρέπει τα παιδιά από να έχουν πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες, σε πολλά διαφορετικά αγαθά και είναι σαφές από την πρώτερη περίοδο προγραμματισμού ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο το δικαίωμα των παιδιών σε ένα αξιοπρεπές βιωτικό επίπεδο και στο ότι θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο στο ότι τα παιδιά δεν θα πρέπει να στερούνται βασικά αγαθά, ότι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όχι μόνο σε επιστημιστική βοήθεια, αλλά και σε υποστήριξη που έχει να κάνει με την υγεία, την εκπαίδευση, τη φροντίδα του και την ε, προστασία τους. Τις ιδέες αυτές έχει προωθήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο στην ε, τελευταία τους ε, τοποθέτηση. Το φαινόμενο λοιπόν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, ιδιαίτερα πολυδιάστατο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η έρευνα που έχει διεξαχθεί δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι τελικά η οικονομική ένδια των γονιών που οδηγεί σε αυτή την πολυδιάστατη ένδια για τα παιδιά. Και τα παιδιά τα οποία ζουν σε ένα τέτοιο φτωχά υλικό περιβάλλον, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να οδηγηθούν σε οικονομική φτώχεια ως ενήλικες. Εμπλέκονται δηλαδή τα παιδιά σε ένα φαύλο κύκλο, σε μια μακροχρόνια δηλαδή διαδικασία παιδικής φτώχειας, που εν συνεχεία γίνεται οικονομική φτώχεια όταν γίνουν τα παιδιά αυτά ενήλικες. Τον κύκλο αυτό τον φαύλο θέλουμε εμείς να σπάσουμε με την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε πώς έχει κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παιδική φτώχεια. Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε για την καταμέτρηση παιδική φτώχεια δεν είναι πλέον ιδανικά, γιατί ουσιαστικά μετράμε περισσότερο εδώ πέρα τη φτώχεια των οικοκυριών και έπειτα ενσωματώνουμε και τα παιδιά σε αυτούς τους δείκτες. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας ξεχωριστός, αν θέλετε, δείκτης. Όταν βλέπουμε λοιπόν τα γενικά αυτά αριθμητικά δεδομένα που βλέπετε στη διαφάνεια, βλέπουμε ότι πάνω από το 25% των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν έτη 2016 βρισκόντουσαν στο όριο της φτώχειας και κινδύνευαν από κοινωνικό αποκλεισμό. Και κάτι που είναι ακόμα πιο σημαντικό, 8 εκατομμύρια από αυτό το 25% βρισκόντουσαν σε καθεστώς ε, σοβαρής στέρησης ε, σημαντικών αγαθών και υπηρεσιών φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε οριζόντια σε πολλά Σε ορισμένα βέβαια εκδηλώνεται με τρόπο ιδιαίτερα σοβαρό. Η γραφική αυτή παράσταση, μόνο ότι δεν μπορεί να διαβάσετε ακριβώς, καταδεικνύει τελικά τις πολλές διαφορετικές αυτές πτυχές του κινδύνου της ε, φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Και με κόκκινο βλέπετε όλες αυτές τις περιπτώσεις όπου έχουμε εντοπίσει σοβαρές υλικές στερήσεις. Και βέβαια έχουμε και περιπτώσεις ε, όπως η Σουηδία και το Λουξεμβούργο που βρισκόμαστε κάτω από το 1% ενώ έχουμε και περιπτώσεις όπως την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα όπου το ποσοστό αυξάνεται πολύ σημαντικά. Σαφώς δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα είναι οξύ και αν θέλετε και η όλη δυναμική είναι εντελώ διαφορετική. Ο συνολικός αριθμός των ε, παιδιών που κινδυνεύουν από φτώχεια παρουσιάζει μείωση την τελευταία δεκαετία, αλλά αν δούμε επιμέρους τα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 κράτη-μέλη, στα οποία είχαμε μάλιστα και αύξηση. Πώς ανταποκρινόμαστε στο πρόβλημα αυτό μέσω συγκεκριμένων πολιτικών. Πρόβλημα που, όπως σας είπα, παραμένει ιδιαίτερα οξύ και παρουσιάζει και αύξηση ορισμένα κράτη-μέλη. Σαφώς μπορούμε να πούμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο Υπάρχει μια γενικότερη συνένεση ότι θα πρέπει να γίνουν απαραίτητε επενδύσει για να σπάσει αυτό ο φαύλο κύκλο τη παιδική φτώχεια και ότι θα πρέπει να καταφέρουμε τελικά να επενδύσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσουμε τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς να αντιμετωπίσουν την ένδυα αυτή. Μάλιστα σε συστάσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια τη νομοθετικής αυτή περίοδου, αλλά και από συστάσει και ψηφίσματα που είδαμε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπουμε ότι υπάρχει η πρόθεση αυτή. Υπάρχει λοιπόν γενικότερη συνένεση για τις επενδύσεις αυτές, ωστόσο όταν εξετάζουμε τα επιμέρους εθνικά στρατηγικά πλαίσια, αν δούμε τις προτεραιότητες στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, βλέπουμε ότι δεν επικεντρωνόμαστε παρκώς το ζήτημα της παιδικής φτώχειας, ότι δεν έχουμε επενδύσει ή προγράμματα τα οποία να καταπολεμούν ειδικά το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας. Υπάρχουν εθνικά προγράμματα που αναλύουν το πρόβλημα αυτό, αλλά ο αριθμός των ειδικών αναχώρα συστάσεων που έχουν να κάνουν με την παιδική φτώχεια παρουσιάζει μείωση από 7 το 2014 σε 0 πέρσι. Επομένως, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αρκετά ισχυρή βούληση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών για το ζήτημα αυτό. Αναλύσαμε έπειτα τη χρηματοδότηση από συγκεκριμένα ταμεία. Μα ενδιαφέρει εδώ ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Ευρωπαϊκή Βοήθεια στου Απόρου, το ΦΕΑΝΤ. Στο ΦΕΑΝΤ υπάρχουν συγκεκριμένοι δείκτε, ισχύουν συγκεκριμένε προποθέσει στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού η ε, καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και η κοινωνική ενσωμάτωση έχουν προωθηθεί περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, αλλά και πάλι δεν έχουμε προγράμματα που να έχουν να κάνουν ε, αποκλειστικά και μόνο με την παιδική φτώχεια. Ή προγράμματα που να έχουν να κάνουν ε, με παιδιά τα οποία στερούνται βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά κατά νου, η δική μας μελέτη προσπάθησε να εντοπίσει χρηματοδοτικές παρεμβάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν ως τελικό αποδέκτη κυρίως τα παιδιά και τα μειονεκτούντα παιδιά, τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν, πλήττονται από σοβαρές υλικέ στερήσεις. Βλέπουμε εδώ πέρα, σε σχέση με τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά, ότι υπάρχουν πλέον συγκεκριμένοι τομείς από τα τρία αυτά προγράμματα που βλέπετε στη διαφάνεια, που έχουν να κάνουν με την παιδική φτώχεια. Για παράδειγμα, το Ταμείο Ευρωπαϊκή Βοήθεια στου Απόρου το ΦΕΑΤ προβλέπει ε, επισητιστική και ηλική βοήθεια, καθώ επίση και προγράμματα κοινωνική ενσωμάτωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μα δίνει ακόμα περισσότερε δυνατότητε. Έχουμε προγράμματα που έχουν να κάνουν με ποιοτική φροντίδα των παιδιών. Ιδίω ε, για τις περιοχές εκείνες που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια πιο έντονη γεωγραφική συγκέντρωση ε, σε συγκεκριμένε περιοχέ, οι οποίε πλήττονται όλου ιδιαίτερω. Έχουμε προγράμματα που έχουν να κάνουν ε, με, την, ε, με τις προσβάσιμες υπηρεσίες εκπαίδευσης, έχουμε άλλα προγράμματα που αφορούν την κοινωνική στέγαση και που δίνουν προτεραιότητα κυρίως στα νοικοκυριά εκείνα τα οποία έχουν παιδιά, τα οποία πλήττονται από φτώχεια. Βλέπετε αυτά τα μέτρα, καθώς επίσης και άλλα μέτρα, τα οποία πλέον προβάλλονται πολύ περισσότερο σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, σε επίπεδο παρέμβασης. Αν δούμε τώρα την πιο σφαιρική συνολική εικόνα, πώς δηλαδή χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη την κοινωνική χρηματοδότηση προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Έχουμε ένα τέταρτο των πόρων του ESF που προβλέπεται για μέτρα κοινωνικής ενσωμάτωσης, 8 δισεκατομμύρια για παράδειγμα έχουν να κάνουν με προγράμματα καταπολέμησης της πρόορης εγκατάλειψης του σχολείου. Παρ' όλα αυτά δεν είμαστε σε θέση από τα δεδομένα τα οποία έχουμε σε κοινωνικό επίπεδο να δούμε πραγματικά ποια είναι τα ποσά τα οποία δίδονται ειδικά για το στόχο της καταπολέμησης τη ε, παιδική φτώχεια. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτά με τα εφιστάμενα διοικητικά δεδομένα. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα στα πλαίσια του ΦΕΑ, του Ταμείου Ευρωπαϊκή Βοήθεια στου Απόρου. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι εκεί πέρα τα πράγματα παρουσιάζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια. Βλέπουμε όντω ποια είναι τα προγράμματα εκείνα τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ως απότερο στόχο τα παιδιά εκείνα τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρές ηλικέ στερήσεις. Αλλά βλέπετε ότι και σε άλλα προγράμματα έχουμε για παράδειγμα 6 δισεκατομμύρια τα οποία δίδονται για την εκπαίδευση, ένα εκατομμύριο δίδεται συγκεκριμένα για την προσχολική εκπαίδευση και ξέρουμε μέσω ερευνών που έχουμε κάνει ότι η προσχολική επίσης εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα προκειμένου να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της παιδικής φτώχειας. Εν γέννη βλέπουμε ότι για το ΦΕΑ, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους, καταφέρνουμε να έχουμε ως αποδέκτες 11 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως μέσω της επισητιστικής βοήθειας. Πολύ μικρότερο είναι το ποσοστό εκείνο των παιδιών το οποίο υποφελούνται ε, στο πλαίσιο προγραμμάτων ηλική ε, υποστήριξη και βλέπουμε πάλι ότι τα παιδιά αυτά εντοπίζονται σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά, Η υποστήριξη αυτή είναι σαφώς αποτελεσματική στην πράξη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Όπως σας είπα, η γενική εικόνα δεν είναι αρκετά σαφής. Τα κράτη-μέλη κάνουν συγκεκριμένες επενδύσεις στον τομέα της παιδικής φτώχειας, ιδίως ε, στα προγράμματα εκείνα που έχουν να κάνουν με την πρόορια εγκατάλειψη του σχολείου ή με την προσχολική παιδεία. Λιγότερες, όμως, είναι επενδύσει που γίνονται στις ε, υγειονομικές η άλλες κοινωνικές υπηρεσίες βρίσκονται σε άλλους τομείς, όπως όλα αυτά, από ΑΠΟ ή Ιδρυματοποίηση μελέτε που κάναμε συγκεκριμένε αυτα απο τις μελέτες που καναμε συγκεκριμενε χώρες, μολονότι μπορεί να μην είναι πολύ συγκεκριμένη η σφαιρική αυτή εικόνα, υπάρχουν παρόλα αυτά συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο, εκεί που υπάρχει ένα συγκεκριμένο εθνικό επενδυτικό πλαίσιο μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση παιδική φτώχεια, Εκεί όντω χρησιμοποιούνται από τα κράτη αυτά πάρα πολύ αποτελεσματικά οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Ευρωπαϊκή Βοήθεια στους Απόρου. Βλέπουμε για παράδειγμα μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία στην Πολωνία, χάρη στην οποία περισσότερα παιδιά είχαν πρόσβαση στην προσχολική παιδεία, ιδίω στι αγροτικέ περιοχέ. Έχοντας κατά νου λοιπόν αυτή τη σφαιρική εικόνα, θα ήθελα τώρα να περάσω γρήγορα στις, στα συμπεράσματα και τις συστάσεις που κάνουμε στη μελέτη μας. Όσον αφορά την επερχόμενη περίοδο προγραμματισμού, εξετάσαμε την υφιστάμενη πρόταση και βλέπουμε ότι τώρα εντοπίζουμε καλύτερα την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας ως στόχο, σαφή ξεκάθαρο ξεχωριστό στόχο για τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και έχουμε πλέον και νέες ευκαιρίες τις οποίες θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε, θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε και συγκεκριμένα να απαιτήσουμε, όπως προβλέπετε, από τα κράτη-μέλη να έχουν συγκεκριμένες στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας, για την κοινωνική ενσωμάτωση και προβλέπετε ότι στη θέσπιση αυτής της εθνικής στρατηγικής θα πρέπει να υπάρχουν και μια συγκεκριμένη καταμέτρηση της α, παιδικής φτώχειας. Και όσον αφορά την εξάντερη σημότητα που ίσχυε για την υφιστάμενη περίοδο προγραμματισμού, και εκεί προβλεπόταν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν το εθνικό πλαίσιο πολιτική για τα ζητήματα αυτά. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις νέε αυτές ευκαιρίες, τις νέες αυτές απαιτήσει ουσιαστικά που προβάλλονται για τα κράτη-μέλη, προκειμένου να προβληθεί περισσότερο ο στόχος της καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας για τα κράτη-μέλη και ιδίω τα κράτη-μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν πιο έντονα προβλήματα, όπως φάνηκε στα στατιστικά δεδομένα τα οποία σας παρουσίασα. Μια σημαντική ευκαιρία που μας δίνεται αυτή τη στιγμή είναι να θέσουμε για τα κράτη-μέλη ένα συγκεκριμένο στόχο που έχει να κάνει με συγκεκριμένε πτυχές παιδικής φτώχειας. Ξέρετε ότι όταν μπορούμε και καταμετρούμε κάτι πιο εύκολα το αντιμετωπίζουμε. Μία άλλη ευκαιρία που μας δίδεται με τη νέα περίοδο προγραμματισμού είναι να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν πιο έντονα προβλήματα να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την παροχή υπηρεσιών ειδικά για παιδιά. Και θα πρέπει τα κράτη αυτά μέλη να μπορούν να εντοπίσουν συγκεκριμένε περιφέρειες στην επικράτειά του, οι οποίε θα μπορέσουν να αποφεληθούν από μια τέτοια χρηματοδότηση. Οι χώρε οι οποίε κατάφεραν τα πάνε καλά στην τρέχουσα και σε προηγούμενε περιόδου προγραμματισμού είναι τα κράτη-μέλη εκείνα που κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν συγκεκριμένε περιφέρειε, συγκεκριμένε γεωγραφικέ ζώνε, στι οποίε θεώρησαν ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητε επενδύσει. Είναι τελικά σε τέτοια κράτη-μέλη, τα οποία είχαν την προσέγγιση αυτή, που καταφέραμε τελικά να βοηθήσουμε περισσότερα παιδιά. Μπορούμε επίση να έχουμε και πιο συγκεκριμένε κατηγορίε παρέμβαση και μπορούμε επίσης να επεκτείνουμε περισσότερο τους δείκτες εκείνους που καλύπτουν ε, τα παιδιά κάτω των 18 στο σύνολο των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ουσιαστικά εμεί αυτό το οποίο εκτιμούμε είναι ότι α, ε, ακόμα και αν γίνει κάτι τέτοιο δεν θα δημιουργηθεί υπερβάλλον διοικητικό άχθος και ακόμα και αν συμβεί κάτι τέτοιο, ακόμα και αν δηλαδή δημιουργήσουμε περαιτέρω διοικητικό φόρτο σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως αξίζει να κάνουμε κάτι τέτοιο γιατί θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση των παιδιών σε όλους τους τομείς πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ευχαριστώ πολύ. Όντω είναι από τα θέματα που έχουν ε, ενδιαφέρον για την Επιτροπή μας και που δείχνει και ευαισθησία για την παιδική φτώχεια. Ευχαριστώ. Τελευταία η ομιλήτρια είναι η κυρία Κάλμα η οποία θα μας μιλήσει για άλλο σημαντικό θέμα που είναι η διεθνή συνεργασία και η διασυνοριακή. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τρία σημεία θα δανειστώ από τον προλαλήσαντα και θα σας δώσω κάποια στοιχεία και κάποια σχόλια βάσει της εργασίας που έχει γίνει από το, την αντίστοιχη πλατφόρμα την υπερεθνική η ESF ε, που διαχειρίζεται το ε, ε, EID που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενημέρωση και την τοπική ανάπτυξη. Η Μανουέλα Σάμεκ μίλησε για τη σημασία της ενίσχυσης και της διατήρησης της εταιρική σχέσης στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Είναι σημαντικές αυτές οι εταιρικέ σχέσεις για να αντιμετωπίζουμε περίπλοκες καταστάσεις και προβλήματα που καλύτερα να αντιμετωπίσει και να λύσει και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η εταιρική σχέση είναι πολύ σημαντική, διδάσκεται ο ένας από άλλον, η δημόσια διοίκηση, οι διαχειριστικές αρχές, διάφορα επίπεδα συνεργάζονται με τους δικαιούχους, είτε είναι ΜΚΟ, είτε είναι κοινωνική εταιρή, είτε άλλοι. Έτσι, μαθαίνει ο ένας από τον άλλον. Υπάρχει μια άλλη υποστήριξη. Να σας δώσω δύο επιτυχή ε, παραδείγματα από τη συγκεκριμένη υπερεθνική πλατφόρμα. Φλάνδρα. Εδώ στο Βέλγιο η Φλάνδρα είναι διαχειριστική αρχή που έχει συμπεριλάβει όλους τους δικαιούχους και τους αρμόδιους φορείς σε όλα τα προγράμματα ε, από την αρχή της, τη σχεδίαση, την υλοποίηση, την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ε, συζητούν με τους διάφορους δικαιούχους και ενδιαφερομένους τις ανάγκες, ας πούμε, της φλαμαδικής αγοράς εργασίας και πώς μπορεί να αναλυφθεί συγκεκριμένη δράση για να βελτιώσει τα επιχειρησιακά προγράμματα. Επίσης, οι δικαιούχοι καλούνται και οι ενδιαφερόμενοι να αξιολογήσουν τα προγράμματα. Γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις ε, από την προκήρυξη του διαγωνισμού ακόμα, δηλαδή πριν προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός και μια ε, ε, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, έχουν λόγο οι ενδιαφερόμενοι οι stakeholders. Επίσης, ε, διοργανώνουν ε, επισκέψεις στα έργα, συνεχείς και τακτικές και προωθούν ε, την δημιουργία εταιρικών σχέσεων σε τοπικό επίπεδο. Άλλο παράδειγμα που θεωρώ επίσης ε, ε, σημαντικό και σχετικό είναι αυτό της Βουλγαρίας. Στη Βουλγαρία έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδο στα τελευταία χρόνια σε, από ιδρυματοποίηση, όπως αναφέραμε προηγουμένως και για την παιδική φτώχεια. Το γεγονός όμως ότι το Εθνικό Δίκτυο για τα παιδιά συμμετείχε ε, σε ε, επιτροπές παρακολούθησης και ελέγχου θέθη ως συγκεκριμένο στόχος στη συμφωνία εταιρική σχέσης αυτή η αποϊδρυματοποίηση. Και επίσης βρέθηκαν και τα απαραίτητα κονδύλια που δόθηκαν για τη δημιουργία δυνατοτήτων και ικανοτήτων των ΜΚΙΟ. Τι δείχνουν αυτά τα δύο επιτυχή παραδείγματα, ότι οι εταιρικέ σχέσεις όταν σχεδιάζονται και εφαρμόζονται σωστά μπορούν να συνεισφέρουν και ε, στην ενίσχυση της δημιουργίας ικανοτήτων και για τις δημόσιες διοικήσεις αλλά και για τους ίδιους τους ενεχομένους. Ένα δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτό της ε, παιδικής φτώχειας και ιδιαίτερα η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης συμφωνώ πάρα πολύ με τον Χάρολτ Μπροτσάιτης για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο δεν έχει ασχοληθεί αυτή την προγραμματική περίοδο με τα παιδιά ως συγκεκριμένη ομάδα στόχου. Έτσι χάθηκαν ευκαιρίες στη χρήση ε, των πόρων από το ΕΚΤ για να αντιμετωπιστεί η παιδική φτώχεια. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η νέα πρόταση ε, το ESF Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ρητά τα παιδιά ως ομάδα στόχο της χρηματοδότησης και όχι μόνο αυτό, υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο που έχει σημασία κατά την άποψή μου. Και αυτό αφορά το πώς χρησιμοποιήθηκε το κοινωνικό ταμείο στην καταπολέμηση της φτώχειας και ε, στην κοινωνική ένταξη. Αν δούμε την υλοποίηση και πώς απορροφάται το 20% που αφιερώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, πάνω από το του 25% μάλιστα ε, έχει δαπανηθεί για την ενεργή ένταξη και κυρίως την ενεργή ένταξη ε, στην αγορά εργασίας. Εμείς τι πιστεύουμε. Η νέα πρόταση ESF Plus συμπεριλαμβάνει λοιπόν την καταπολέμηση της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού ως ξεχωριστό στόχο, ανεξάρτητο της απασχόλησης. Καθώς επίσης και το γεγονός ότι αναφέρονται ρητά τα παιδιά ως ομάδα στόχος, αυτά τα δύο στοιχεία ε, ελπίζουμε να βοηθήσουν και να οδηγήσουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο σε απορρόφηση του 25% του ΕΚΤ, ακριβώς για να λυθούν τα προβλήματα και να βρεθούν τα μέτρα αντιμετώπισης κάποιων ε, ε, ομάδων του πληθυσμού που είναι εκτός αγοράς εργασίας, όπως είναι τα παιδιά, ηλικιωμένοι ή ανίκανοι προς εργασία. Άλλο σημαντικό σημείο, η μείωση της φτώχειας θα πρέπει επίσης να αποσυνδεθεί, να απαγκιστρωθεί από τον κοινωνικό ε, αποκλεισμό και την καταπολέμηση του. Άλλο παράδειγμα, η αποϊδρυματοποίηση υπάρχει σε διάφορα κράτη-μέλη και όχι μόνο στα κράτη-μέλη όπου υπάρχει η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα. Άρα, στο μέλλον ε, θα μπορούσε να υπάρχει μια σύσταση που να λέει σύμφωνα με τον κανονισμό περί γενικών διατάξεων, να υπάρχουν αυτές ε, οι πρόνοιες σε όλα τα κράτη-μέλη και να υπάρχουν και στρατηγικές. Όχι απλώ γενικώ εκρίζωση της στόχιας και της παιδικής, αλλά η ε, κοινωνική ένταξη να είναι ο στόχος. Ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να αναφέρω έχει να κάνει με την ε, διοικητική δυνατότητα και τις ικανότητες των ε, δημοσίων διοικήσεων, τον έφερε ο καθηγητής Σάντορ. Συμφωνώ απολύτως ότι η ενίσχυση των εθνικών διοικήσεων σε διάφορα επίπεδα και των δυνατοτήτων τους είναι εκ των για να είναι αποτελεσματική όσο και παραγωγική η ε, απορρόφηση των κονδυλίων. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή ε, των μελών και των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θεματικό στόχο 11 που αφορά την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στο ESF+. Θα βρείτε άλλες διατάξεις για τη δημιουργία δυνατοτήτων των ενδιαφερομένων κτλ. Αλλά η διοικητική μεταρρύθμιση είναι κάτι που ε, μεταφέρεται στο πρόγραμμα υποστήριξης των διαφθορτικών μεταρρυθμίσεων, σε άλλο πρόγραμμα δηλαδή, ε, και, όπου δεν είναι αρμόδια η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Άρα, εμείς θα συστήναμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό, πώς θα γίνει ε, ο συντονισμός των διαφόρων μέσων και εργαλείων έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχουν καλύτερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων μέσων. Γιατί η διοικητική ικανότητα ενός κρατικού μηχανισμού έχει πολύ μεγάλη σημασία για να υλοποιούνται κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι του ESF+, όπως είναι ο εξχρονισμός των υπηρεσιών και μεταξύ αυτών και των υπηρεσιών ε, των δημοσίων ε, Βελτίωση βελτίωσης της εκπαίδευσης και τη κατάρτιση των εργαζομένων, βελτίωση στην πρόσβαση στην υγεία και στα συστήματα κοινωνική ασφάλισης που και αυτά χρειάζονται εξυγχρονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους εμπειρογνώμονες. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρουσίαση αυτή και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να μιλάμε και ζητώ συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά ξέρουμε ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο για τη διερμηνία. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Εγώ ως εισηγήτρια θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Αν και με ενδιαφέρει να ακούσω περισσότερα εσάς παρά να μιλάω εγώ. Μας βοηθάνε πάρα πολύ αυτά που μας λέτε. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με την απορρόφηση των κονδυλίων, ιδιαίτερα εκείνων που ε, στοχεύουν στην καταπολέμηση της ε, ανεργίας των νέων. Γίνεται μέγας λόγος για αυτό το θέμα και κυριαρχεί και στο Κοινοβούλιο η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Αλλά επειδή τα κράτη-μέλη έχουν ε, δυσκολίες να βρουν τους εθνικούς πόρους για να καταπολεμήσουν την ανεργία των νέων και αναφέρθηκε και ο καθηγητής Άντορ, έχει εγκριθεί η εμπροστοβαρής εκταμίευση, οι προκαταβολές. Και επίσης δεν χρειάζεται εθνική συγχρηματοδότηση. Με τη νέα πρόταση ε, ε, των κοινών διατάξεων μειώνεται η συγχρηματοδότηση των κρατών μελών και ουσιαστικά ε, όμως εξαφανίζεται η προκαταβολή, η εμπροστοβαρής χρηματοδότηση, το front loading αυτό πώς θα επηρεάσει ε, την υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανεργία αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και τα μεγαλύτερα ε, προβλήματα για να εκταμιεύουν ε, τα ποσά αυτά εκ των προτέρων. Και δεύτερη ερώτηση αφορά το Ταμείο Βοήθειας στους Απόρους μιλούμε για συγχώνευση των ταμείων και όλοι συμφωνούμε ότι αυτό θα βοηθήσει και το ΦΕΑΤ και το ESF ε, να ε, συγχωνευθούν καλύτερα για να υπάρχει καλύτερη υποστήριξη και ηλική και να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Μας λένε όμως ότι οι κοινωνικές ε, υπηρεσίες ότι κινδυνεύουν να διαλυθούν αυτοί οι στόχοι μέσα στο γενικό σύνολο και να χαθούν. Ακραία φτώχεια υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη, αυτό μας το είπαν συνάδελφοι και ο κύριος Μάν μεταξύ άλλων. Άρα ε, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί αυτή η βοήθεια στους απόρους για να φτάνει στους πλέον ε, πληγέντες. Πώς θα σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της φτώχειας για να έχουν όλη την ευκαιρία να βγουν από τη φτώχεια αυτή. Αυτά και σταματώ εδώ γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικές και εκτενέστατες οι παρουσιάσεις σας και σας ευχαριστώ και πάλι. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο και να κάνει κάποιες ερωτήσεις στους εμπειρογνώμονες. Σε Έχετε το λόγο. Κύριε Άντορ, πρώτο. few comments and θα ξεκινήσω με μερικά σχόλια. Σίγουρα οι συνάδελφοι θα συμπληρώσουν. Είναι κρίσιμα τα ερωτήματα. Για την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, ο τρόπος που διευθετείται η χρηματοδότηση θα πρέπει να συσχετίζεται με την μακροοικονομική κατάσταση και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ανεργία των νέων ανταποκρίνεται στους κύκλους ε, των επιχειρήσεων. Αυξάνεται η ανεργία όταν ε, μειώνεται η οικονομία και ταυτόχρονα όταν ε, το κράτος μέλος έχει πιο σοβαρούς περιορισμούς παρά σε κανονικούς καιρούς. Και αυτό εξηγεί και την ανάγκη για την προχρηματοδότηση που έχει εισαχθεί από το, 2000, από το 2015. Με συγχωρείτε. Άρα, κατά την άποψή μου, τότε, εάν είναι μέσα ή εκτός του ESF, αυτό δεν είναι το κρίσιμο ερώτημα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ότι θα πρέπει να ε, γνωρίζουμε ποιος είναι ο κύκλος, ο οικονομικός και πώς είναι αυτός ο κύκλος και ε, η ανάγκη για αυτού του τύπου ε, παρέμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντατικότερη και εντονότερη όταν ένα κράτος μέλος έχει ε, λιγότερο ε, χώρο ε, δημοσιονομικής κίνησης. Τώρα, σχετικά με το ΤΕΒΑ, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους, είναι πιο περίπλοκο το ερώτημα, διότι λέτε πώς θα σπάσουμε τον φαύλο θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στην πρόληψη. Θέματα, για παράδειγμα, που αφορούν τους άστεγους. Είναι πιο εύκολο να προλάβουμε την στέγης και την κλιμάκωση των προβλημάτων σε κάποια κράτη-μέλη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, είχαν μειώσει το ποσοστό των αστέγων σε μεγάλο βαθμό. Τώρα από την ε, κρίση έχει επιταχυνθεί και ενταθεί το πρόβλημα. Οι Ευρωπαίοι μετανάστες που συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες υπάρχει και το θέμα της υπευθυνότητας της όταν ένας δήμος δεν αισθάνεται αρμόδιος ε, για ε, την αύξηση των μεταναστών και αγνοεί αυτή την πτυχή και αυτό οδηγεί στην αύξηση των δαπανών. Όμως αυτό είναι θέμα για παράδειγμα το θέμα των Ρωμά, ιδιαίτερα στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια, το εάν θα ανεχτούμε την συγκέντρωση της ηλικής ε, στέρησης ε, που παρατηρείται εκεί και αυτό που είδαμε το 10 και το 11 όταν ήμουν υπεύθυνο για την ένταξη των Ρωμά, χωρίς παρέμβαση, ισχυρή παρέμβαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή καθοδήγηση πολιτική και χρηματοδότηση, το εθνικό επίπεδο ποτέ δεν θα ε, προβεί σε επαρκή δράση. Ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σάμεκ. Θέλετε να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια. Να κάνω εγώ Θα κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις, ιδίως όσον αφορά τους νέους. Ο οικονομικός κύκλος και η κρίση είναι σίγουρα ένας παράγοντας και σίγουρα η ενεργεία των νέων είναι υψηλότερη εκεί που ισχύουν οι πιο δεινοί, αν θέλετε, οι πιο δεινές οικονομικές συνθήκες. Έχει να κάνει όμως και με την ρύθμιση της αγοράς εργασίας ή με τις πολιτικές εκείνες που έχουν να κάνουν με τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην, ή από το Πανεπιστήμιο στον χώρο εργασία. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολύ θετικά διδάγματα από τις χώρες εκείνες που έχουν εφαρμόσει επιτυχή προγράμματα. Μπορούμε να δούμε δηλαδή τι έχει γίνει σε συγκεκριμένε περιστάσεις και συνθήκες. Έχουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πρόορια εγκατάλειψη του σχολείου, ζήτημα το οποίο θίχτηκε σε προηγούμενη παρουσίαση. Ξέρετε ότι έχουμε ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν ένα υψηλό ποσοστό νέων και οι οποίοι είναι άεργοι, ουσιαστικά δεν ψάχνουν καν για εργασία. Και ξέρετε ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες, κυρίως οι νέες γυναίκες, που πλήττονται από το φαινόμενο αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να διοχετεύσουμε πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές σε τέτοιες ομάδες. Το ζήτημα της προχρηματοδότησης συνδέεται προφανώς με την οικονομική κρίση, συνδέεται με την δημοσιονομική δυσπραγία. Συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή. Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα όσον αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους. Πάντως, για τις πιο μειονεκτούσες ομάδες, σαφώς θα πρέπει να έχουμε νέες μορφές παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο. Να καταφέρουμε να συνδυάσουμε διαφορετικές μορφές υποστήριξης, επιστηστική βοήθεια, υποστήριξη όσον αφορά τη στέγαση, αλλά και νέες υπηρεσίες έβρασης εργασίας. Το να ομαδοποιηθούν, αν θέλετε, οι παρεμβάσεις αυτές στα πλαίσια ενό ταμείου είναι θετικό, ενδεχομένω να μην είναι πολύ εύκολο στην αρχή να διαχειριστούμε με ένα ομοιογενή τρόπο όλα αυτά τα προγράμματα, προκειμένου δικαιούχοι να μπορούν πραγματικά να συμμετέχουν περισσότερο σε ένα ταμείο το οποίο θα είναι τελικά πολύ πιο πολύπλευρο ή το οποίο θα, θα χρηματοδοτεί πολλές διαφορετικές δράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Μπρουζάητης. Σύντομα, πάρα πολύ. Θέλω να προσθέσω κάτι στο τελευταίο. Και στις δικές μας μελέτες βλέπουμε ότι ένας τρόπος ολοκλήρωσης των υπηρεσιών είναι η προώθηση αυτής της εδαφικής διάστασης. Πράγμα που γίνεται αυτή την προγραμματική περίοδο με τις επενδύσεις. Δηλαδή, οι ντόπιες κοινωνίες γνωρίζουν περισσότερο τα προβλήματα και τις προκλήσεις τους και έτσι με συντονισμένο τρόπο και με συνεργασία με τις τοπικές αρχές εκτελείται και το ε, ε, Κοινωνικό Ταμείο. Ε, ευχαριστώ η κυρία Κάιμα. Σε ό,τι αφορά το ΤΕΒΑ, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους πόρους ΦΕΑΤ, είναι πολύ σημαντικό φυσικά να έχουμε επιστημιστική βοήθεια και υλική βοήθεια προς τους πόρους, τους όσοι υποφέρουν από υλικές στερήσεις. Θα πρέπει όμως ε, να πάμε και παραπέρα, όχι απλώς να τους δίνουμε τρόφιμα και κάποια υλική βοήθεια. Να προχωρήσουμε και σε πολιτικές πρόληψεις γιατί το να δίνεις ε, τροφή και συσίτια ε, μπορεί να σώσει κάποιον που βρίσκεται στη φτώχεια προσωρινά, αλλά δεν χειραφετεί το φτωχό, δεν τον βοηθάει να βγει από τη φτώχεια, διαιωνίζεται η κατάστασή του. Πολύ λίγα είναι τα κράτη-μέλη που αποφάσισαν να συνδυάσουν τα δύο επιχειρησιακά προγράμματα, πράγμα που επιτρέπεται στο σημερινό ΤΕΒΑ. Το πιο αποτελεσματικό μέτρο εδώ θα ήταν ακριβώς αυτό, να συνδεθεί η ηλική βοήθεια με τα μέτρα για την κοινωνική ένταξη. Ευχαριστώ πολύ τους ε, εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς προφανώς, όπως πάντα. Είμαστε ευγνώμονες για τη δουλειά τους και οι διερμηνείς ευχαριστούν την πρώτη. Λήξη συνεδρίασης. Μέχρι τις 16 του Σεπτέμβρη, δεν απατώ, με σε 9 το πρωί. Στις 6 Σεπτέμβρη, συγγνώμη. Α, όχι, στις 10 μου λένε, 10 και μισή, όχι 9, έχει αλλάξει η ώρα. Ωραία, λοιπόν. 6 του μηνός Σεπτεμβρίου στις 10.30 συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ.